good, morning everybody. Καλημέρα λοιπόν κυρίες και κύριοι. Ο Μέγαν Καντίκ. Θα μιλήσω ουγγρικά. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους. Καλωσορίζουμε και τον καθηγητή Ντόναλτ Μπρομ από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ θα ξεκινήσει με μία παρουσίαση. Δίνουμε το λόγο στον καθηγητή Μπρουμ. Sorry, number two, number two is English. yes. Thank you. Thank you very much, Chairman. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για την καλή μεταχείριση των ζώων και θα ξεκινήσω με κάποιους όρους. Θα μιλήσω για την υγεία, για την ευαισθησία, για την επιρροή της πρόσφατης πολιτικής και νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως στον τομέα της μεταχείρισης των ζώων και επίσης θα μιλήσω και για κάποιες ευκαιρίες για ευρωπαϊκές εταιρείες ως αποτέλεσμα της πολιτικής και νομοθεσίας για την ε, ορθή μεταχείριση των ζώων, για τις ε, εξαγωγές των Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και επίσης θα αναφερθώ στο πώς χρησιμοποιούνται κάποιοι όροι στην νομοθεσία, κάποιοι επιστημονικοί όροι για νομοθεσία που αφορά συγκεκριμένα τα ζώα και όταν αναφέρεται η ορθή διαβίωση των ζώων σε άλλου είδους νομοθεσία, παραδείγματος χάρη στην εμπορική νομοθεσία. Θα σας πω και δύο λόγια για τους αριθμούς, για τον πληθυσμό των ζώων, για το τι καλύπτεται από νομοθεσία και τι όχι και τέλος για το τι απαιτείται ως νομοθεσία για την ορθή μεταχείριση των ζώων, κάποια στοιχεία επιστημονικά και στοιχεία για προγράμματα εκπαίδευσης και η ορθή διαβίωση των ζώων είναι τμήμα της βιωσιμότητας και πτυχή της βιωσιμότητας. Ένα παραγωγικό σύστημα μπορεί να είναι μη βιώσιμο όταν έχει ανεπιθύμητες ενέργειες στην ανθρώπινη υγεία. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται συζητήσεις σχετικά με τα, σύστημα και με τα συστήματα ε, ιατρικής και κτηνιατρικής ε, πρακτικής μεταξύ άλλων που μπορούν να προκαλούν αυξημένη αντιμικροβιακή αντίσταση και επομένως να έχει επίπτωση στην ε, περίθαλψη των ανθρώπων και των ζώων. Μπορεί να έχει επιπτώσεις επίσης στην ε, διαβίωση των ζώων, ε, η γενετική τροποποίηση για μεγάλο μέρος του πληθυσμού μπορεί να είναι μη αποδεκτό ή να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες. Επιζήμια επίπτωση στο περιβάλλον επίσης μπορεί να οδηγεί σε αλλαγή του κλίματος ή να επηρεάζει τη βιοπικιλότητα ή να προκαλεί ρήπανση. Μπορεί επίσης να μην χρησιμοποιούνται σωστά οι παγκόσμιοι επισητιστικοί πόροι μία οι αποδοτικές πρακτικές μπορεί να μην είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα. Όταν δίνουμε λοιπόν στα ψάρια ως τροφή, τροφή που προέρχεται από ηχθείς, δεν είναι εξίσου βιώσιμο όσο αν τους δίναμε ε, τροφή που προέρχεται από φυτά. Επίσης, ε, ε, στα, ε, στις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες, το 90% των τροφών που δίδονται είναι τροφές που δίδεται, δίδονται και σε ανθρώπους. Θα, μπορούσαμε λοιπόν, θα μπορούσαμε να δίνουμε διαφορετικού είδους τροφή, λοιπόν, για την καλύτερη χρήση των πόρων παγκοσμίω. Επίσης, υπάρχουν και θέματα δίκαιου εμπορίου, δηλαδή πολλοί δεν θέλουν να αγοράσουν καφέ όταν ο καφές παράγεται από εργαζομένους που αμείβονται ελάχιστα και όλο το κέρδος πηγαίνει στις εταιρείες ε, που εκμεταλλεύονται τους εργαζομένους και παράγουν τον καφέ. Το δίκαιο εμπόριο λοιπόν είναι μια έννοια που επηρεάζει τους πολίτες και το επιθεμητό είναι η παραγωγή, ιδίως στις πιο φτωχές χώρες, να αμείβονται επαρκώς για αυτό το οποίο παράγουν. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι οι αγροτικές κοινότητες και η διατήρηση αυτών και η επιβίωσή τους. Και αυτό είναι ένας παράγον που μπορεί να κάνει ένα σύστημα μη βιώσιμο. Βάζω λοιπόν και την ορθή διαβίωση των ζώων μέσα σε αυτό το σύστημα. Υπάρχουν πολλοί τομείς και ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι τομείς ε, που απασχολούν την Επιτροπή σας. Σας είπα λοιπόν ε, πώς ένα σύστημα μπορεί να είναι μη βιώσιμο. Οι παράγοντες αυτοί όμως αποτελούν ε, και ένα τμήμα της κρίσης των πολιτών για τα προϊόντα για την ποιότητα των ειδών διατροφής. Η ποιότητα εξαρτάται από τη γεύση και από τη θρεπτική του αξία, αλλά και από τον τρόπο παραγωγής. Δηλαδή, οι πολίτες ταξινομούν ένα, ε, μια τροφή ως κακής ποιότητας αν έχει αρνητική επίπτωση σε κάποιους από τους τομείς βιωσιμότητας που προανέφερα. Υπάρχει η έννοια της ε, ορθής διαβίωσης των ζώων των οργανισμών. Η όρος ορθή διαβίωση χρησιμοποιείται και για τους ανθρώπους, όχι μόνο για τα ζώα, αλλά δεν χρησιμοποιείται για τα φυτά ή για τα άψυχα αντικείμενα. Άρα η διαβίωση ενός ατόμου είναι η κατάστασή του όσον αφορά την προσπάθειά του να επιβιώσει στο περιβάλλον του. Πρέπει να κατανοήσουμε τις ανάγκες ε, διαβίωσης ορισμένων ε, ζώων των οργανισμών. Πρέπει να δούμε τι είναι σημαντικό για τα ζώα και τι τους συμβαίνει αν δεν τους εξασφαλίζονται κάποιοι βασικοί πόροι. Επίσης μπορούμε να σκεφτούμε στοιχεία που επηρεάζουν ε, την διαβίωση, οι ορμόνες παραδείγματος χάρη, η μεταφορά ε, τα πρόβατα παραδείγματο χάρη ε, εκρίνουν κάποιε ορμόνε. και αν φορτώσει ένα κοπάδι πρόβατα ε, σε ένα φορτηγό ε, αρχίζουν να εκρίνουν ορμόνες διότι βρίσκονται σε κατάσταση επίγουσα ανάγκη σε ένα άγνωστο περιβάλλον προσαρμόζονται μετά από 48 ώρες αν τα ζώα ταξιδεύουν σε αυτοκινητόδρομο πέφτει ε, το επίπεδο των ορμονών, αλλά αν μετά περάσει το φορτηγό σε ένα δρόμο με πολλές στροφές ε, και συνεχίζει ο οδηγός να ε, οδηγεί γρήγορα στις στροφές, η κορτιζόλη που εκρίνει το, το ζώο αυξάνεται και πάλι γιατί βρίσκεται σε κατάσταση μη αναγνωρίσιμη. Μία πρόσφατη μελέτη στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ εξετάζει τον πόνο στα πρόβατα. Μπορεί να κάνεις γκριμάτσες όταν ε, πονάς, ε, να σφίγγεις το πρόσωπό σου, να κλείνεις τα μάτια. Αυτό που κάνει το μωράκι που βλέπετε στην ε, φωτογραφία το κάνουν και άλλα ζώα και τα ποντίκια και τα πρόβατα και τα άλογα και μπορεί το επίπεδο του πόνου στα ζώα να προσδιοριστεί και από αυτή την απόκριση υπομορφή γκριμάτσας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως ε, σημείο αναγνώρισης του πόνου για την αναγνώριση ασθένειας ή κακής μεταχείρισης. Η ορθή διαβίωση των ζώων λοιπόν αναφέρεται σε όλους τους μηχανισμούς που επιστρατεύει ένα ζώο για να ανταποκριθεί στο περιβάλλον του, φυσιολογικούς, ε, συμπεριφορικούς, ε, καθώς και αισθήματα και ανταπόκριση στην παθολογία. Μπορεί να έχει θετικά αισθήματα, αρνητικά αισθήματα. Η έννοια της υγείας ε, έχει άμεση σχέση για την ε, ορθή διαβίωση των ζώων και η υγεία είναι βασικό κομμάτι της ε, καλής διαβίωσης. Δεν είναι χωριστό. Η υγεία είναι η κατάσταση του ατόμου που έχει σχέση με την παθολογία και προσπαθεί να αντιμετωπίσει κάθε παθολογία. Η ορθή διαβίωση είναι ευρύτερος όρος, άρα η υγεία είναι μία πτυχή της ορθής διαβίωσης. Κάποιοι από τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται εδώ είναι πεπαλαιωμένοι. Ο ορισμός του, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, παραδείγματος χάρη, είναι απριχαιωμένος. Η διαβίωση λοιπόν είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των ζώων. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την ε, διαβίωση ε, ενός πληθυσμού γενικότερα, μόνο κατά μέσο όρο η προστασία των ζώων είναι κάτι το οποίο κάνουν οι άνθρωποι. Ενώ η διαβίωση είναι κάτι το οποίο κάνει το ζώο. Υπάρχουν νόμοι αυτή τη στιγμή που περιορίζονται όμως για ορισμένα ζώα και συνήθως περιορίζονται στα ζώα τα οποία θεωρούνται ευαίσθητα. Ευαισθησία για τα ζώα σημαίνει ότι, σημαίνει ότι ε, έχει την επίγνωση και την γνωστική ικανότητα ώστε να έχει αισθήματα. Να υπάρχει δηλαδή εγκεφαλική λειτουργία για θετικά και αρνητικά αισθήματα όπως ο, φόν, ο φόβος, ο πόνος, η ευχαρίστηση. Συνήθως προστατεύουμε τα ευαίσθητα ζώα περισσότερο από τα ζώα που δεν είναι ευαίσθητα. Θα μπορούσε να πει κανείς ποιοι άνθρωποι είναι ευαίσθητοι. Αν σκεφτείτε ένα ε, ανθρώπινο οάριο που έχει γονιμοποιηθεί, αναπτύσσεται σε έμβριο, αναπτύσσεται στο εσωτερικό της μητέρας και τελικά γεννάται ως μωρό. Αυτό το άτομο που γεννάται, το μωράκι, είναι ευαίσθητο, έχει αυτή την έννοια που αποκαλούμε ευαισθησία, δεν την έχει όμως ως έμβριο. Και δεν είναι ευαίσθητα όλα τα ζώα. Επίσης υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ε, κάποια εγκεφαλική βλάβη και δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της ευαισθησίας. Τα επιστημονικά δεδομένα μας δείχνουν ότι τα θηλαστικά, τα πτηνά, τα ερπετά, τα αμφίβια, οι ηχθείς ε, και ορισμένα άλλα ζώα, κεφαλόποδα, χταπόδι, καλαμάρι, σουπιά, ε, καθώς και καβούρια, αστακοί, γαρίδες είναι ευαίσθητα. Και άλλα ζώα μπορούμε να προσθέσουμε, προς το παρόν αυτά έχουμε στον κατάλογό μας. Άλλος ένας όρος που χρησιμοποιείται είναι η ποιότητα ζωής. ποιότητα ζωής σημαίνει ορθή διαβίωση, σημαίνει το ίδιο πράγμα, αλλά χρησιμοποιούμε την ποιότητα ζωής για αυτά τα οποία διαρκούν για περιορισμένο διάστημα. Δεν μιλάμε για κακή ποιότητα ζωής αν κόψουμε το δάχτυλό μας, αλλά ε, έχουμε λιγότερο καλή διαβίωση αν έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Οι όροι καλή διαβίωση και υγεία έχουν το ίδιο νόημα και για τους ανθρώπους και για τα άλλα ζώα. Δεν υπάρχει διαφορά. Και μας ενδιαφέρει η κοινή υγεία και ε, διαβίωση ανθρωπίνων όντων και άλλων ζώντων οργανισμών. Όταν ε, η ε, ορθή διαβίωση ενός ατόμου δεν είναι επαρκής, ανταποκρίνεται με διαφορετικό τρόπο στις ασθένειες, επομένως αν βελτιώσουμε την διαβίωση, μειώνουμε και τις ασθένειες η πρόληψη της αντιμικροβιακής αντίστασης είναι θετική για την καλή διαβίωση και αν βελτιώσουμε την διαβίωση έχουμε καλύτερο νοσοποιητικό σύστημα, επομένως έχουμε μικρότερη ανάγκη για αντιμικροβιακά προϊόντα. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τόσα φάρμακα όταν έχουμε καλή διαβίωση στην εκτροφή των ε, ζώων. Είναι σημαντικό λοιπόν να τονίσουμε αυτούς τους όρους. Ένας άλλος όρος είναι η ευθανασία τον όρο αυτό πρέπει να το χρησιμοποιούμε κατά τον ίδιο τρόπο για ανθρώπους και άλλα ζώντα ζώα. Ευθανασία σημαίνει ε, ότι θανατώνεται ένα άτομο προς όφελος του ιδίου ατόμου με τρόπο ε, ανθρωπιστικά ορθό. Εάν ωφελείται κάποιος άλλος δεν πρέπει να ονομάζεται ευθανασία, πρέπει να ονομάζεται θανάτωση θανάτωση με ανθρωπιστικό τρόπο, αλλά όχι ευθανασία. Εάν έχουμε λοιπόν ένα κατοικίδιο ζώο και δεν ε, ε, ε, θέλουμε να το κρατήσουμε και το θανατώσουμε, δεν, ανα... δεν το αποκαλούμε ευθανασία, το αποκαλούμε θανάτωση, ακόμη και αν το κάνουμε με ανθρωπιστικά ορθό τρόπο. Η φροντίδα λοιπόν για τους ανθρώπους και η φροντίδα για τα ζώα από τους ανθρώπους δίδεται κατά καλύτερο τρόπο εάν θεωρούμε και τους ανθρώπους και τα ζώα ως άτομα. Αν έχουμε λοιπόν 10.000 κοτόπουλα και τα μεταχειριζόμαστε σαν να ήταν ζώντα ζώα ίσης αξίας με τον άνθρωπο, θα, θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Η διαβίωση εκατοντάδων χιλιάδων ζώων έχει βελτιωθεί από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ορθή διαβίωση των ζώων. Αυτό είναι το συμπέρασμα από τη μελέτη μου. Και σε άλλα μέρη του κόσμου όμως έχει βελτιωθεί, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχει βελτιωθεί λόγω των πολιτικών και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νομοθεσία λοιπόν σε άλλες χώρες συχνά έχει αντιγράψει ε, στοιχεία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ε, και χρησιμοποιεί ευρωπαϊκή νομοθεσία ή εκθέσεις του ΕΦΣΑ ε, ή άλλων οργανισμών, παραδείγματος χάρη η έκθεση για τα θηλυκά γουρούνια που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και χρησιμοποιηθεί και σε άλλα μέρη του κόσμου για να αποφευχθούν οι απάνθρωπες μέθοδοι εκτροφής θηλυκών γουρουνιών. Ε, η πολιτική λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ορθή διαβίωση των ζώων, ε, καθώς και η νομοθεσία, έχει θετικές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτό τον τομέα, νομοθεσία δηλαδή για την ορθή διαβίωση, ε, σε αυτό τον τομέα η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει βελτιωθεί διότι θεωρείται δείκτης πολιτισμένης κοινωνίας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς προέκυψε αυτή η θετική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία από τις αλλαγές που επέφερε νέα νομοθεσία στην, για τη διαβίωση των ζώων και έχει κάνει και το κοινό να δει τέτοια νομοθεσία, είναι η βελτίωση των γνώσεων για τα ζώα, ανησυχούν περισσότερο και ενδιαφέρονται περισσότερο σε πολλές χώρες οι πολίτες για τη διαβίωση των ζώων. Η έρευνα, καθώς και η επιβολή του νόμου και τα προγράμματα εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν περαιτέρω προωθήσει αυτή την θετική ανάπτυξη. Και ήταν σημαντική επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα μέρη του κόσμου. Από ευρωπαϊκές έρευνες είναι σαφές ότι οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχούν για τη διαβίωση των ζώων όχι μόνο αν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τα ζώα που δεν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυξάνεται αυτή η τάση τα τελευταία 20-30 χρόνια σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο μια ευρωπαϊκή τάση, ισχύει και σε άλλα μέρη του κόσμου. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολιτική βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία όπως τις εκθέσεις του ΕΦΣΑ και σε στοιχεία από μελέτες οι οποίες είναι, οι οποίες είναι πολύ καλά διαρθρωμένες όπως οι εκθέσεις του ε, Ευρωβαρομέτρου. Η απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προϊόντα φώκιας νομοθετήθηκε λόγω επιστημονικών δεδομένων που έδειχναν ότι οι μέθοδοι θανάτωσης των νεαρών ζώων ήταν απάνθρωπες. Η ευζοία των ζώων και η ορθή μεταχείριση αναφέρεται από πολλές οργανώσεις παγκοσμίως. Η ΦΑΟ λέει ότι η ορθή διαβίωση των ζώων θεωρείται ότι έχει το δυναμικό να δημιουργήσει ωφέλη και για τους παραγωγούς και για τα εκτρεφόμενα ζώα. Η Παγκόσμια Οργάνωση Επιζωτιών έχει ε, ε, Εκδόσεις συστάσεις για διάφορα θέματα στα οποία έχουν συμφωνήσει 185 χώρες. Ο ΩΣΑ έχει πολιτικές για την ορθή διαβίωση των ζώων, η Διεθνής Χρηματοοικονομική Εταιρεία, η IFC, τμήμα της Παγκόσμιας Τράπεζας, δηλώνει ότι τα καλύτερα πρότυπα για την διαβίωση των ζώων βελτιώνουν την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και την κερδοφορία ικανοποιούν τις διεθνείς αγορές και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών. Υπάρχουν ε, λοιπόν ευκαιρίε ε, για τι ε, εταιρείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω αποτέλεσμα τη πολιτική για την καλή διαβίωση των ζώων. Γενικά, αν κάποιο είναι ο πρώτο που κάνει κάτι στον κόσμο, έχει και τις περισσότερες ευκαιρίε. Και νομίζω ότι αυτό σε κάποιο βαθμό ισχύει. Δεν θα έλεγα ότι πρόκειται για μια τεράστια αγορά, είναι όμω αρκετά σημαντική. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη σφαγή των ζώων οδήγησε στην ανάπτυξη μεθόδων για την αναισθητοποίηση και διαχείριση των ζώων, πρώτα σε χώρες που ήθελαν να εξάγουν τα προϊόντα τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατόπιν σε άλλες χώρες που ανέπτυξαν ε, νομοθεσία για την ε, σφαγή με ανθρώπινα κριτήρια. Ε, σε σφαγεία λοιπόν στην Κίνα για παράδειγμα χρησιμοποιούνται προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποια σφαγεία. Τα έχω δει και εγώ ίδιος. Εάν λοιπόν έχει κανείς ε, καλό σύστημα ανεστοποίησης ε, και εσφαγής, μπορεί ε, να πωλήσει κανείς τον εξοπλισμό αυτόν. Επίσης, πολλούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και συστήματα και εξοπλισμός για διάφορα άλλα προϊόντα που συνδέονται με την κτηνοτροφία. Υπάρχουν ευκαιρίες και για την πώληση προϊόντων για την καλή διαβίωση των ζώων. Εάν λοιπόν σκεφτούμε τον ΠΟΕ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, δεν καθορίζει την καλή διαβίωση των ζώων ως λόγο για περιορισμό των εισαγωγών. Και αυτό, όπως γνωρίζετε, έχει δημιουργήσει προβλήματα ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απαγόρευση προϊόντων φώκιας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υιοθετήθηκε επειδή θεωρήθηκε ότι ο τρόπος που σκοτώνονται οι φώκες αυτές δεν είναι ανθρώπινος είτε τα σκοτώνουν στο ξύλο, τις ε, μικρές φώκες, ε, είτε τις ε, πυροβολούν. Η φώκια βρίσκεται πάνω σε ένα κομμάτι πάγου που πλέει και δεν σκοτώνεται πάντα αμέσω η φώκια. Το ίδιο ισχύει όταν τις σκοτώνουν στο ξύλο. Δεν πεθαίνει πάντα αμέσω η φώκια. Υπήρχαν λοιπόν καλά επιστημονικά στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται και σε μια έκθεση της ΕΦΣΑ που έδειχναν ότι ο τρόπος που σκοτώνονταν οι φώκες δεν ήταν πάντα ανθρώπινος και το ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θεωρούσαν ότι είναι λογικό να απολύεται ένα προϊόν όταν ε, το προϊόν προέρχεται από το δέρμα ζώου που, σκοτώθηκε, που ε, ε, το χωτάρανε ενώ, ενώ είχε ακόμα τις αισθήσει του. Και αυτό ε, παρουσιάστηκε ως θέμα δημόσιας ηθικής, ε, μια υπεράσπιση την οποία τελικά δέχτηκε ο ΠΟΕ. Κάτι που μπορεί να οδηγήσει και σε, άλλες, ε, σε άλλους περιορισμούς εισαγωγών λόγω δημόσιας ηθικής, διότι η δημόσια ηθική αναφέρεται από τον ΠΟΕ ως λόγο για τον περιορισμό της κυκλοφορίας προϊόντων. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρονται τα ευαίσθητα ζώα και η καλή διαβίωση των ζώων σε νόμους που σχετίζονται και με το εμπόριο. Ε, από την συνθήκη του Άμστερνταμ και τη συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρονται τα ζώα ως ευαίσθητα ε, όντα, ενώ άλλα νομοθετήματα αναφέρονται στα ζώα ως αντικείμενα ή ιδιοκτησία. Έχουμε και εμείς, για παράδειγμα, την ε, οδηγία για την προστασία των ζώων όταν χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, όπου αναφέρεται ότι τα ζώα έχουν μία αξία την οποία θα πρέπει να σεβόμαστε. Πρέπει πάντα να τα μεταχειριζόμαστε ως ε, ευαίσθητα όντα. Υπάρχει εδώ λοιπόν ε, σαφής ε, αναφορά ε, στις ε, αισθήσεις του ζώου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν γίνεται αυτό. Για παράδειγμα, στην συμφωνία ΣΥΤΑ με τον Καναδά δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να αναφέρονται τέτοιες διατάξεις σε, σε περισσότερα νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περισσότερες συμφωνίες. Επίσης, αυτή τη στιγμή η οδηγία 9859 λέει ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαβίωση των ζώων, θα πρέπει να διασφαλίζεται η καλή διαβίωση των ζώων, ε, διότι πρέπει να τηρούνται κάποια επίπεδα. Επίσης, οι ανάγκες ε, είναι κάτι, ε, είναι μια λειτουργία του εγκεφάλου, είναι λοιπόν βιολογικές οι ανάγκες, όχι φυσιολογικές, όχι σωματικές ή συμπεριφοριστικές τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο και τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δούμε τα ζώα που ε, έχει ο κόσμος ε, στην Ευρώπη, το πιο ε, σύνηθες ζώο είναι το κοτόπουλο, 4, ε, δισεκατομμύρια και το, στη δεύτερη και τρίτη θέση βρίσκονται η Πέστροφα και ο Σολομός, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο είναι άλλα είδη. Κατόπιν έχουμε κότες, κουνέλια, πάπιες, ε, γαλοπούλες, ε, γουρούνια, γάτες, ε, βοηδοί, πρόβατα και σκυλιά. Και κατόπιν έχουμε ζώα εργαστηρίου και άλλα είδη, τα οποία δεν λέω ότι δεν είναι τόσο σημαντικά, είναι όμως λιγότερα. Και αν υπάρχει πρόβλημα ε, καλής διαβίωσης, ε, τότε είναι πολύ πιο πιθανό να... Το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο αν πρόκειται για κοτόπουλο ή για ψάρι ηχθειοτροφείο. Έχουμε νομοθεσία για τα ζώα για επιστημονική χρήση όσον αφορά την ε, μεταφορά και σφαγή των ζώων, τα ζώα σε ζωολογικούς κήπους. Έχουμε επίσης κανόνες ε, για ε, κοτόπουλα, βοηδή, ε, χείρους κλπ. Το πρόβλημα όμως είναι ότι το τέταρτο κατά σειρά, πέμπτο, όγδο, δέκατο και ενδέκατο ζώο που έχουν οι άνθρωποι στην κατοχή τους δεν καλύπτονται από την νομοθεσία. Καλύπτεται η στέγαση των ζώων και η σφαγή, αλλά το, η μεγαλύτερη διάρκεια τη ζωή του, όταν δεν μεταφέρονται ή όταν δεν σφάζονται, δεν καλύπτονται οι συνθήκε διαβίωση των ζώων αυτών, εκτός από την οδηγία 9858, που όμως έχει τόσο γενική διατύπωση, που μάλλον ε, έχει πολύ περιορισμένα αποτελέσματα. Ποια είναι λοιπόν τα προβλήματα αυτά. Τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι τα προβλήματα των ποδιών στα κοτόπουλα ε, για κρεατοπαραγωγή. Και τώρα που έχουμε νομοθεσία για τις οτόκες όρνηθες, ε, τους χείρους ε, και τα βοηδή, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι γαλακτοφόρες αγελάδες. Ε, δεν καλύπτονται και συχνά υποφέρουν από παράλυση, μαστίτιδα και αναπαραγωγικά προβλήματα. Ε, μάλιστα σε ποσοστό 30 με 40% των ε, ατόμων. Είναι σημαντικά τα προβλήματα αυτά ε, για τα ζώα. Η παραγωγή γάλακτος λοιπόν δημιουργεί σημαντικά προβλήματα για τα ζώα και ιδιαίτερα τα πιο παραγωγικά είδη. Είναι λοιπόν πρόβλημα το ότι δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία. Έχουμε νομοθεσία για την υγεία των ζώων που υιοθετήθηκε πρόσφατα. Οι περισσότεροι πολίτες Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θεωρούν απαράδεκτο ότι 300 εκατομμύρια ζώα, ε, ψάρια ηχθειοτροφίου, πέστροφα σολομό, ε, καθώ και κουνέλια, πάπιε γαλοπούλες, αγελάδες, χείρι, σκύλοι και γάτες δεν καλύπτονται από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια κράτη-μέλη έχουν σχετική νομοθεσία, άλλα όχι. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν μπορούν να φερθούν από άνθρωπα και νόμιμα ε, σε τέτοια ζώα σε κάποια κράτη-μέλη. <clears throat> Και ε, κάποιες ε, τρίτες χώρες ε, γελάνε μαζί μας για το λόγο αυτό. Αν είχαμε λοιπόν έναν γενικό νόμο για την προστασία των ζώων, θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε όλα τα ζώα αυτά. Και επίσης θα μπορούσαμε να έχουμε τμήματα της νομοθεσίας για τα ή ξεχωριστά νομοθετήματα για τα βασικά είδη θα έπρεπε να αναφέρεται η καλή διαβίωση των ζώων και η ευαισθησία των ζώων σε συμφωνίες εμπορικές και άλλη νομοθεσία που να μην ε, αναφέρεται συγκεκριμένα στα ζώα, αλλά που μπορεί να καλύπτει ζώα σε κάποιο βαθμό. Τι μελλοντική δράση απαιτείται λοιπόν. Νομίζω ότι ε, οι ευκαιρίες για εκπαίδευση όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων είναι ε, πολύ σημαντική και αναφυσβήτητα. Ο καλύτερος τρόπος να γίνει κάτι τέτοιο είναι μέσω διαδικτύου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε κάποιες περιπτώσεις ε, έχει παράσχει πολύ καλή πληροφόρηση μέσω διαδικτύου. Αυτή τη στιγμή όμως δεν γίνεται στο συγκεκριμένο τομέα αυτό. Είχαμε το τους δείκτες για την καλή διαβίωση των ζώων, ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντό τη εντολή του προγράμματο αυτού συμπεριλαμβανόταν η δημιουργία ε, μιας ιστοσελίδας ε, για την ε, εκπαίδευση στην καλή διαβίωση των ζώων. Αυτό έγινε, αλλά δεν συνεχίζεται και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια ή κάποια παρόμοια και θα πρέπει να παρέχεται χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να παρέχονται επιστημονικά στοιχεία υψηλής ποιότητας και να παρέχεται εκπαίδευση για την διαβίωση των ζώων σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται θα πρέπει να πρόκειται για αντικειμενικές πληροφορίες επιστημονικά βάσιμες. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πληροφορίες προς ανθρώπους με συγκεκριμένα συμφέροντα ε, που μπορεί να είναι χρήσιμες, αλλά δεν είναι ε, αμερόληπτες πληροφορίες αυτές και δεν, είναι αντικειμενικές και δεν έχουν στηριχθεί επιστημονικά. Επίσης, θα πρέπει να συνεχιστούν οι πολιτικές σε κάποιες χώρες που έχουν αποδείξει την αξία τους. Ακόμα βρισκόμαστε σε θέση όπου χρειαζόμαστε περισσότερους δείκτες για την καλή διαβίωση των ζώων σε συγκεκριμένους ε, τομείς. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερες επιστημονικές έρευνες πάνω στο θέμα αυτό. Χρειαζόμαστε μελέτες και χρειαζόμαστε και μελέτες σχετικά με τα αποτελέσματα των δικτών για την καλή διαβίωση των ζώων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράδειγμα από έναν ε, κτηνίατρο επιθεωρητή ή ε, από ε, έναν κτηνοτρόφο για να ελέγξει την καλή διαβίωση των ζώων του. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε καλύτερα την καλή διαβίωση των ζώων με άλλους παράγοντες σε συστήματα βιώσιμα, διότι ο συνδυασμός αυτών αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων η πολιτική των ε, ελέγχων και της ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή και εδώ και κάποιο καιρό είναι πολύτιμη και θα πρέπει να συνεχιστεί. Πιστεύω όμως ότι η επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ε, συμπλήρωση της νομοθεσίας. Πρέπει να έχουμε καλή επιβολή. Αυτό όμως δεν λύνει όλα τα προβλήματα, διότι υπάρχουν πολλά κενά δεν μπορεί κανείς να ε, εφαρμόσει νομοθεσία που δεν υπάρχει. Πρέπει λοιπόν ε, να έχουμε νομοθεσία και να εφαρμόζεται σωστά. Βλέπετε τώρα τον ε, τίτλο της μελέτης, καθώς και δύο ακόμα βιβλία που έχω συγγράψει πάνω στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Τμήμα Πολιτικής και τον Εκτάβια Μαζόκη και τους συναδέλφους του που με βοήθησαν στην εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Mr. Professor, thank you indeed. Ευχαριστούμε κυρία καθηγητά. Εγώ είμαι βιοχημικός και μου είναι ιδιαίτερα προσφυλή αυτά τα οποία είπατε. Άκουσα την παρουσίασή σας με μεγάλη προσοχή. Μια πολύ χρήσιμη παρουσίαση για όλους μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε ερωτήσεις για τον καθηγητή Μπρούμ. Παρακαλώ. Ε, ε, Okay, Gentlemen. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, όποιος θέλει ας έχει το λόγο. Η κυρία Χάσενκαπ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε ευγενέστατοι εδώ. Όλο ένας παραχωρεί στον άλλο τη θέση του για την πρώτη ερώτηση. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το συζητάμε πολύ συχνά. Συνήθως στο Κοινοβούλιο μιλάμε για τους ανθρώπους και μάλιστα για τους ανθρώπους της δύση και κυρίως για τα χρήματα των ανθρώπων που ζουν στη Δύση. Είναι σημαντικό να μιλάμε ένα ολόκληρο πρωινό για την ορθή διαβίωση των ζώων και θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Και καλό θα ήταν να θεσπίσουμε ε, καλύτερη νομοθεσία για τα ζώα που το αξίζουν. Έχω δύο ερωτήσει προς τον καθηγητή Μπρούμ. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή Αναφορών ε, που έθεσε αυτό το σημαντικό θέμα και ευχαριστώ τον καθηγητή Μπρούμ για την παρουσίαση αυτής της πολύ σημαντικής μελέτης Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη ε, θεωρεί ότι έχει τα υψηλότερα πρότυπα για την ορθή διαβίωση των ζώων στον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, ξέρουμε ότι εκτρέφονται ζώα σε βιομηχανικές ε, εγκαταστάσεις. Ξέρουμε ότι καταλυστεύονται οι θάλασσες. Βασανίζουμε φρικτά τα ζώα. Διάβασα σε έκθεση ότι πετάνε ε, γαϊδούρια από υψηλά κτίρια. Νόμιζα το χειρότερο που είχα δει στην Ευρώπη ήταν ότι έκαιγαν ταύρου, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν και χειρότερα. Πάντα με εκπλήσουν ε, τα άκρα στα οποία μπορεί να φτάσει η κακία του ανθρώπου έναντι των ζώων. Όσον αφορά τώρα την νομοθεσία για την μεταχείριση των ζώων, κύριε καθηγητά, νομίζετε ότι αν διατηρήσουμε την ισχύουσα αναστολή το μορατόριο που ισχύει τα τελευταία χρόνια θα χάσουμε την πρώτη θέση για την ευζοία των ζώων. Άλλες χώρες θα μας ξεπεράσουν, η Βραζιλία, η Ινδία, η Κίνα. μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε ότι έχουμε τα υψηλότερα πρότυπα για την διαβίωση των ζώων στον κόσμο ή πρέπει να θεσπίσουμε νέα νομοθεσία για να κρατήσουμε τα πρωτεία. Στην παρουσίασή σας μιλήσατε για τη βιωσιμότητα και για το τι είναι βιώσιμο και τι όχι. Μιλήσατε και για το δίκαιο εμπόριο, για δίκαιη μεταχείριση των παραγωγών στις φτωχές χώρες. Στην Ευρώπη βλέπουμε, στα σούπερ μάρκετ παραδείγματο χάρη, εδώ στην πλατεία απ' έξω από το κοινοβούλιο, στην πλατεία του Λουξεμβούργου, βλέπουμε ότι ένα λίτρο γάλα κοστίζει 29 λεπτά του ευρώ. Το δίκαιο εμπόριο και η βιωσιμότητα θα έπρεπε να καλύπτουν το εμπόριο και στην Ευρώπη που δεν είναι τόσο φτωχές οι χώρες μας, αλλά θα έπρεπε να είναι δίκαιη η πολιτική και για τους δικούς μας αγρότες. Γιατί το να πουλάμε ένα λίτρο γάλα 29 λεπτά του ευρώ, νομίζω ότι είναι κλοπή και δεν είναι καθόλου δίκαιο. Ευχαριστώ πολύ. Θα συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις για τον καθηγητή Μπρούμ για να απαντήσει όλες μαζί. Ο κύριος Εκ. Θα μιλήσω γερμανικά, την μητρική μου γλώσσα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Μπρούμ για την πολύ καλή αυτή μελέτη, την εξαιρετική αυτή μελέτη, διότι έτσι στρέφει το ενδιαφέρον στο θέμα της καλής διαβίωσης των ζώων. Το μόνο που θα ήθελα να επικρίνω στην μελέτη αυτή ήταν ε, οι τελικές παρατηρήσεις. Φυσικά, κύριε Μπρούμ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει κάποιες προόδους στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων. Αλλά, δεδομένου του πόσο υποφέρουν τα ζώα, οι, ε, οι πρόοδοι αυτές είναι ε, περιθωριακές. Ε, δεκάδες εκατομμύρια χιλιάδες εκατομμύρια κοτόπουλα σκοτώνονται μόνο και μόνο επειδή είναι αρσενικά. 55 εκατομμύρια ε, κοτόπουλα τον χρόνο μόνο και μόνο επειδή είναι αρσενικά και δεν μπορούν να γεννήσουν αυγά. Είναι απίστευτο το τι γίνεται στον τομέα της κτηνοτροφίας σφαγή των ζώων ε, χωρίς ε, επαρκή αναισθητοποίηση. Πρόκειται για τεράστια καταστροφή, για τεράστιο σκάνδαλο. Η κονικλοτροφία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έλαβε, υιοθέτησε σχετική πρόταση την προηγούμενη εβδομάδα. Στα 60 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν εξετάσουμε πώς η νομοθεσία έχουμε υιοθετήσει στον τομέα της ε, καλής διαβίωσης των ζώων, με μεγάλα γράμματα θα χωρέσουν όλα τα νομοθετήματα σε μία σελίδα α4. Ενώ αν κοιτάξετε άλλους τομείς ε, μπορούμε να ε, συμπληρώσουμε τόμους βιβλίων. Και όλοι το λένε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενδιαφέρεται για προτάσεις για την καλή διαβίωση των την προστασία των ζώων. Ο κύριος Ιούνκερ και ο κύριος Τίμερμαν λίγο πολύ το έχουν πει επίσημα ότι κατά τη διάρκεια της δικής τους θητείας δεν θα εκδοθεί νέα πρόταση για την προστασία των ζώων. Ε, και έχουμε ένα πολύ ε, χοντρό παράδειγμα το οποίο εμένα με έχει συγκλονίσει. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά, πολλά είδη ζώων, όπως είπε ο κύριος Μπρούμ, που δεν καλύπτονται από την νομοθεσία. 330 ε, εκατομμύρια ε, κουνέλια τον χρόνο εκτρέφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σφάζονται το χρόνο, που ζουν σε κλουβιά που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό των ζώων αυτών. Η κονικλοτροφία στην Ευρώπη είναι ε, η, πιο σημαντική νόμιμη μέθοδος ε, βασανισμού των ζώων. Και υπήρξε αντίδραση σε πρότασή μου. Είπαμε ότι θέλουμε βελτίωση της κατάστασης. Θέλουμε να υιοθετηθεί νομοθεσία για ένα είδος ζώου που επί 60 χρόνια το... δεν είχαμε ασχοληθεί καθόλου μαζί του. Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη πριν την ψηφοφορία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι «Α, όχι, αυτό είναι θέμα επικουρικότητας, ε, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Εμείς, ε, λοιπόν, δεν θα αγγίξουμε το θέμα αυτό. Και η Επίτροπος είπε ότι ναι, αν υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από, λόγω πίεσης από ε, μια μη κυβερνητική ομάδα για την προστασία των ζώων, είπε ότι ναι, αν υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον μπορούμε να εξετάσουμε το θέμα. Είναι σκάνδαλο. Είναι απόλυτη αποτυχία των πολιτικών. Από τη μία έχουμε την προστασία των ζώων και από την άλλη έχουμε επιχειρηματικά συμφέροντα. Πάντα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργεί ε, προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων. Το ΕΛΚ επίσης πήρε το ε, ε, μέρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. και αυτά που αναφέρονται για τα κουνέλια ήταν λίγο πολύ αυτά που είχε πει και η Επίτροπος. Κανένα νομοθετικό μέτρο, τίποτα. Όχι, στο μέλλον χρειαζόμαστε πολιτική βούληση για την προστασία των ζώων και τότε θα μπορέσει να γίνει κάτι, τότε θα προσεγγίσουμε τους πολίτες. Οι πολίτες έχουν δείξει ότι θέλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερη προστασία των ζώων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να ε, ακούσει αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό μας εκλέγουν εδώ. Αλλιώς απλά παίζουμε θέατρο και προσποιούμαστε ότι έχουμε δημοκρατία που στην πραγματικότητα δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι το πραγματικό τεστ αυτό είναι το θέμα που θα δείξει πόσο κοντά είναι κοντά στους πολίτες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ακούσει τους πολίτες που ζητάνε καλύτερη διαβίωση των ζώων, ε, κάτι που άλλωστε είναι και θέμα ηθικής. Θα υποβάλει περισσότερες ε, νομοθετικές προτάσεις για την προστασία των ζώων ή θα συνεχίσει όπως τα τελευταία 60 χρόνια. Και μία ε, ερώτηση. Η ερώτησή μου προς εσάς κύριε καθηγητά είναι, πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη την εξαιρετική μελέτη σας στις μελλοντικέ της αποφάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο Πέτερ Γιάρ. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος ΕΚΑ έκανε πολύ καλή εισαγωγή στο θέμα αυτό. Και το μεγαλύτερο μέρος ε, των δηλώσεών του απευθύνονται όχι στον επιστήμονα αλλά σε εμά τους πολιτικούς. Όσον αφορά λοιπόν ε, την ε, καλή διαβίωση των ζώων, υπάρχουν κάποιες οικονομικές πιέσεις, υπάρχει συνένεση στην κοινωνία. Όλα αυτά είναι παράγοντες που διαμορφώνουν την πολιτική. θα μπορούσε να περιγράψει κανείς ε, και πιο θετικά τη συζήτηση για την ε, κονικλοτροφία. Είχαμε μία πρόταση που υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και φυσικά υπάρχει και περιθώριο βελτίωσης. Μπορεί κανείς ε, να κάνει διάφορες δημοσκοπήσεις αλλά ε, υπάρχει και δισταγμός πάντως ε, όσον αφορά τα κουνέλια. Υπάρχει μια σημαντική ε, σύγκρουση στην Ευρώπη. Πάντως το θέμα παραμένει στο θεματολόγιο και η ερώτησή μου προς τον ε, κύριο ε, επιστήμονα είναι η εξή. Φυσικά τη μελέτη δεν ε, θα πρέπει να την κλείσουμε στο σιρτάρι μας, θα πρέπει να την διαδώσουμε. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε μία περίληψη των συμπερασμάτων. Τι θεωρείτε εσείς ότι είναι πιο σημαντικό. Και όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, διεξάγεται δημόσια συζήτηση, ακόμα καθοδόν βρισκόμαστε, αλλά όταν βλέπω πώς μεταχειριζόμασταν τα ζώα πριν 30-40 χρόνια, υπάρχει βελτίωση. Ε, εγώ ξέρω πώς ε, πραγματοποιόταν η κτηνοτροφία στην Ανατολική Γερμανία τότε. Η ερώτησή μου προς εσάς, κύριε καθηγητά, είναι υπάρχει σαφής επιστημονικός ορισμός της καλής διαβίωσης των ζώων. Αυτό θα μας ευκολύνει, διότι θα πούμε ότι να, έχουμε εδώ πέρα μια αντικειμενική βάση. Διότι μερικές φορές αυτό που νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι καλό για τον ζώο μπορεί να διαφέρει από αυτό που αποδεικνύει η επιστήμη. Και επίσης, εσείς πώς βλέπετε την ερασιτεχνική ε, κτηνοτροφία, Δηλαδή μπορεί κάποιο ε, να έχει ένα κουνέλι ως χόμπι. Αυτό πώς το βλέπετε, απαιτείται και εδώ νομοθετική ρύθμιση. Επόμενη ερώτηση. Η στρατηγική μας ε, για την ε, αντιμετώπιση ασθενειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. αντιστοιχεί ε, σε αυτά που θα πρέπει να κάνουμε σύμφωνα με την ε, καλή διαβίωση των ζώων. Επίσης, βλέπετε να υπάρχει σχέση Ε, ανάμεσα στην ε, παραγωγή, την εμπορική παραγωγή των ζώων και την καλή διαβίωση των ζώων. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη μελέτη σας και Χαίρομαι όταν επιστήμονες μπορούν να κάνουν μία σύνοψη για τους πολιτικούς. Είναι χρήσιμο για μας αυτό. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Σέβη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε, κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Μπρούμ για τις μελέτες του και για την ε, ε, μελέτη που μας παρουσίασε σήμερα. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για να δώσουμε νέα πνοή στον αγώνα που κάνουμε, να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε έγκριτους επιστήμονες όπως τον κύριο Μπρούμ. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι και συμφωνώ τους μαζί τους, θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Ωστόσο, είναι ατελής η δράση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και αυτό πρέπει να το διαπιστώσουμε. Δεν γίνεται ουσιαστική δουλειά επιτόπου για την καλή διαβίωση των ζώων. Πρέπει αυτό να το διαπιστώσουμε. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο καθηγητή για τη μελέτη που μας παρουσίασε και ελπίζω ότι όλα αυτά θα χρησιμεύσουν για να ε, δοθεί το εναρκτήριο λάκτισμα έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αναλάβουν πιο σημαντική δράση στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συχνά διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις. Δεν θέλουμε πολύ συχνά να θίξουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την καλή διαβίωση των ζώων. Πρόσφατα, για παράδειγμα, κλείσαμε διάφορες αναφορές που είχαν να κάνουν με τη χρηματοδότηση της εκτροφής ετάβρων για τη συμμετοχή τους σε ε, ταυρομαχίες. Πρόκειται όμως για ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις αυτές και συμμετέχουν οι πολίτες οι οποίοι έχουν υποβάλει σχετικές αναφορές και δυστυχώς τις κλείσαμε πολύ γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση οι Ευρωπαίοι πολίτες μέσω της φορολόγησής τους συμμετέχουν στη χρηματοδότηση της εκτροφής ταύρων που θα χρησιμοποιηθούν για λόγους τραυρομαχιών. Σε κάθε περίπτωση, σε Ε, ε, αδράνησαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπήρξε πλειοψηφία υπέρ της αδράνειας και κλείσαμε τις αναφορές. Και εγώ αυτό το βρίσκω θλιβερό, το βρίσκω δυστυχές και επονίδιστο. Αυτό είναι ένα. Υπάρχουν βέβαια και άλλα θέματα και άλλες αναφορές. Θα μπορούσα για παράδειγμα να σκεφτώ την φαλαινοθυρία Πάρα πολλά θέματα κρύβουμε και τα βάζουμε κάτω από το χαλίδι και δεν θέλουμε να φανούν για να μην ε, μπουν στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια σφαίρα και να μην μιλούμε για αυτά. Θεωρώ ότι πρέπει η καλή διαβίωση των ζώων να ξαναγίνει πολιτική προτεραιότητα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ξανακερδίσουμε μεταξύ άλλων την αξιοπιστία μας έναντι του Ευρωπαίου πολίτη. Ο Ευρωπαίος πολίτη ε, ζητά αλλαγή και αυτό το βλέπουμε παντού ε, σε όλα τα δημόσια φόρουμ και αν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στρέφουν τα νότα του στο πολίτη αυτό είναι κάτι πολύ δυστυχές και θα υπάρξει μεγάλο τίμημα. Θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα. Μιλήσατε για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, τον ΠΟΕ και τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κανείς ε, επιχειρήματα της δημόσιας διοντολογίας σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη απαγόρευση της χρήσης ζωικών παραγόντων προϊόντων, ε, παραγόμενα προϊόντα, υποπροϊόντα δηλαδή, από ζώα που, ε, που βίωσαν πόνο και οδύνη. Σε ποια άλλα φόρουμ θα μπορούσαμε να προβάλλουμε αυτή τη λύση, την τόσο προοδευτική, το πιστεύω, και τόσο σημαντική. Μήπως ε, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιο επιχείρημα στο θέμα το οποίο ε, αυτή τη στιγμή έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας και θα συζητηθεί και έχει συζητηθεί και θα ξανασυζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει να κάνει με το φινικέλαιο το οποίο ε, παράγεται στη Βραζιλία και στην Νοτιοανατολική Ασία και πραγματικά προκαλεί ανυπέρβλητες περιβαλλοντικές καταστροφές και προκαλεί την εξαφάνιση εμφάνιση πολλών ειδών ζώων. Έχουμε ε, το, την κόκκινη λίστα για την ε, προστασία της φύσης από διεθνείς οργανισμούς. Είναι η κόκκινη λίστα, ο κόκκινος κατάλογος με μια σειρά ζώων που διατρέχουν σοβαρό ε, κίνδυνο εξαφάνισης. Για να τα καταπολεμήσουμε όλα αυτά, ενδεχομένω θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το επιχείρημα που αναφέρατε. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να μας δώσετε συστάσεις για το πώς μπορούμε να δράσουμε σε διεθνές επίπεδο στις συναλλαγές και στις συμφωνίες που έχουμε με τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή και συνέπεια σε ό,τι αφορά την καλή διαβίωση των ε, ζώων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος καθηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματά σας. Καταρχάς, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος στον τομέα αυτό. Σε διάφορους τομείς είμαστε πρωτοπόροι παγκοσμίω και αυτό κατέστη δυνατό γιατί ε, άνθρωποι από διαφορετικές χώρες ε, συνεδριάζουν, συναντιόνται, συνενούν και έτσι ε, επιτυχάνουν πράγματα που είναι δύσκολο να επιτύχει μια μικρότερη οικονομική μονάδα. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε πρωτοπόροι οι Ευρωπαίοι στην καλή διαβίωση των ζώων και αν δεν κάνουμε τίποτα τα επόμενα πέντε χρόνια θα χάσουμε αυτή την πρωτιά αφού άλλες χώρες ήδη υιοθετούν νομοθεσία, έξι περίπου χώρες έχουν υιοθετήσει πρόσφατα σχετική νομοθεσία. Αναφερθήκατε ε, στη Βραζιλία, μια χώρα η οποία εξετάζει αυτή τη στιγμή διάφορα νομοθετήματα. Η νομοθεσία που έχει για την προστασία προστασία και διατήρηση της φύσης είναι πολύ πιο μπροστά από την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να κάνουν το ίδιο και να μας ξεπεράσουν και στον τομέα των ζώων. Προς το παρόν καλύπτουν τη χαμένη απόσταση οι Βραζιλιάνοι. Υπάρχουν και άλλες χώρες, η Νέα Ζηλανδία θα πράξει τα δέοντα λίγαν συντόμως από ό,τι φαίνεται. Επομένως απαντώ καταφατικά, ναι, αν δεν πράξουμε τίποτα θα χάσουμε την πρωτιά. Σίγουρα βέβαια κάτι θα κάνουμε. Εάν κάνουμε εκπαιδευτικέ δράσει μόνο, αυτό θα είναι χρήσιμο χρήσιμο. Αλλά ε, θα έχει λιγότερο αντίκτυπο από τον αντίκτυπο που θα μπορούσαμε να έχουμε αν υιοθετήσουμε νέα νομοθεσία σε νέους τομείς. Αναφέρθηκε το θέμα του δίκαιου εμπορίου. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε τους πιο φτωχούς ανθρώπους, τις πιο φτωχές χώρες ως καταναλωτές, εμείς όταν αγοράζουμε κάτι. Και βεβαίως πρέπει να στηρίξουμε και τους Ευρωπαίους γεωργούς και να έχουν μια, ε, μια δίκαιη συμφωνία, ένα καλό deal για παράδειγμα όταν πουλάνε το γάλα τους. Είναι πολύ δύσκολο να τους απαιτούμε να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι καλακτοπαραγωγικές του αγελάδε από τη μία όταν μειώνεται το περιθώριο κέρδους τους από την άλλη και όταν τους πιέζουμε τόσο πολύ με τις τιμές. Τα σούπερ μάρκετ όταν ε, θέλουν να έχουν κράχτη και θέλουν να μειώσουν τη τιμή του γάλακτος και να πουλούν το γάλα σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή για να τραβήξουν καταναλωτές, αν θέλουν να στο πράξουν με ίδιο κόστος, να μην είναι αυτό το κόστος να μην μετακυλίεται στα βάρη του κτηνοτρόφου. Ε, να μην μετακυλίεται το βάρος στους ώμους του κτηνοτρόφου. Είναι, έχουν τεράστια δύναμη τα σούπερ μάρκετ και αυτό πρέπει να υποθεί και να διαχειριστεί ε, να γίνει αντικείμενο διαχείρισης με κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι ένα ευρύτερο ζήτημα το ότι χρησιμοποιούν το προϊόν, το γάλα ως loss leader, έτσι είναι ο όρος στο marketing, ε, ε, ε, ότι δεν θα πρέπει να ε, δέχεσαι τη χασούρα σε ένα προϊόν εσύ ως σούπερ μάρκετ και βεβαίως και να τη μετακυλείς στον παραγωγό σου και να τον, ε, και να τον εξοντώνεις μόνο και μόνο για να τραβήξεις περισσότερους καταναλωτές στο δικό σου μαγαζί οι οποίοι θα καταναλώσουν ποντάρις και πιστεύει τα υπόλοιπα προϊόντα στα οποία θα έχεις μεγάλο περιθώριο κέρδους. Αυτό είναι μια πρακτική που θα πρέπει να υπογραμμιστεί και να αντιμετωπιστεί. Εάν θέλει κανείς να ευθυγραμμιστεί με την επιθυμία των καταναλωτών, ε, τότε πρέπει ως πολιτικός να προχωρήσει παραπέρα. Ε, εάν θέσουμε το ερώτημα στους καταναλωτές, πρέπει να αλλάξουμε τους νόμους για να προστατεύσουμε τα ζώα και να προλάβουμε την κακή διαβίωση των ζώων. Ε, τότε πολύ μεγάλη απάντηση των ερωτώντων θα, απαντήσει, θα είναι καταφατική. Πάρα πολλοί άνθρωποι θα απαντήσουν καταφατικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Δεν θα μπω τώρα σε όλες τις ε, ε, περιοχές και σε όλα τα θέματα. Μιλήσατε για τα πουλερικά, τα οποία μπαίνουν σε ένα μηχάνημα το οποίο λέγεται macerator για να γίνουν shredded chicks, να είναι ε, νεωσή εκτροφής και νομίζουμε ότι είναι το κρέας που χρησιμοποιείται για να κάνει κροκέτες, κοτοκροκέτες. Ε, είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος σαν μέθοδο, γιατί από τη ζωή περνούν στο θάνατο εξαιρετικά γρήγορα τα ζώα αυτά και έτσι υποφέρουν να τον λιγότερο ή και καθόλου με το τόσο ξαφνικό που γίνεται. Η μέθοδος δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ε, τι κάνουμε με αυτά τα ζώα. Δεν θα πρέπει να έχουμε σε συστοιχεία κλωβών χιλιάδες ε, ζώα. Υπάρχουν εναλλακτικές και νομίζω ότι ο κλάδος θα αλλάξει κάποια στιγμή γιατί γνωρίζει πόσο πίεση ασκείται πάνω σε αυτό. Ε, τώρα για την καλή διαβίωση των κουντελιών. Είναι ένα πραγματικά σοβαρό πρόβλημα και κάτι πρέπει να γίνει και μάλιστα πολύ γρήγορα κατά τη γνώμη μου. Μιλήσατε για την πλατφόρμα για την καλή διαβίωση των ζώων. Προσωπικώ πιστεύω ότι είναι πάντοτε καλό να συζητούνται εκτεταμένα όλα αυτά τα ζητήματα. Το ερώτημα όμω που τίθεται είναι ποιο αποτέλεσμα θα έχει αυτή η πλατφόρμα για την καλή διαβίωση των ζώων. Αν δεν έχετε νέα νομοθεσία, η πλατφόρμα αυτή θα έχει μικρά ωφέλη. Χαίρομαι που υπάρχει, την καλωσορίζω, αναρωτιέμαι τι πραγματικά θα κάνει. Και τώρα με ρωτήσατε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη στην έκθεσή μου. Οι φίλοι μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου είπαν ότι τους άρεσε πάρα πολύ που τη διάβασαν, αλλά τα χέρια τους είναι και κάπως δεμένα λόγω πολιτικών που αποφασίζονται σε υψηλότερο επίπεδο. Άρα ε, δεν ε, περιμένω ανυπόμονα να αλλάξουν όλα δραστικά, απλά ελπίζω ότι ένα μικρό πράγμα θα αλλάξει και το πιο σημαντικό είναι να αλλάξουν βεβαίως και οι συνήθειες των καταναλωτών. Όπως είπατε, είναι μεγάλη η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο που πιστεύει ότι κάτι πρέπει να γίνει με την καλή διαβίωση των ζώων. Και η κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι πράγματι κάτι πρέπει να γίνει με την καλή διαβίωση των ζώων. Και εάν η έκθεσή μου μπορεί να συμβάλλει προ αυτή την κατεύθυνση, ήθε. Μακάρι, ευχαρίστω και μακάρι να τη χρησιμοποιήσουν και οι άλλε επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Γεωργία και ούτω καθεξής. Ξέρετε, η επιστήμη για την καλή διαβίωση των ζώων αναπτύχθηκε ε, πολύ γρήγορα. Ο ορισμός που έχω χρησιμοποιήσει έχει προκύψει ε, τελευταία από το ερευνητικό τριών τεσσάρων χιλιάδων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται επιστημονικά στο πεδίο αυτό ε, παγκοσμίω. Ο τρόπος με τον οποίο μιλούν οι επιστήμονες για τα πράγματα δεν είναι ακριβώς ο ίδιος με τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, οι υπόλοιποι άνθρωποι όταν ε, μιλούν για τα ίδια πράγματα. Εξαρτάται αν θα είναι έγγραφο πολιτικής, ένα έγγραφο ενημέρωσης, μια ετικέτα ε, σε ένα προϊόν στο σούπερ μάρκετ πάντοτε θα πρέπει να εδράζεται σε επιστημονικά ε, δεδομένα και για τα κατοικία διαζώα. Μου φαίνεται πολύ περίεργο ότι δεν έχουμε νομοθεσία που να προστατεύει τα σκυλιά και τις γάτες όταν ε, οι περισσότεροι άνθρωποι με τα χειρίζονται με τα σκυλιά και τις γάτες τους καλύτερα από τα ζώα εκτροφής, αλλά υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει καθόλου καλή διαβίωση των ζώων αυτών. Δεν είχαμε τέτοια νομοθεσία γιατί θεωρήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ε, πρέπει να υπάρξει νομοθεσία μόνο για τα ζώα τα οποία αποτελούν αντικείμενο ευρέω εμπορίου και γι' αυτό αυτά τα ζώα μπήκαν στην νομοθεσία προστασίας ενώ τα κατοικίδια ζώα, ζώα συντροφιά δεν είναι αντικείμενο ευρέω εμπορίου και γι' αυτό δεν μπήκαν στην νομοθεσία. Αυτό είναι δηλαδή φυσική απόρρια του τρόπου με τον οποίο κινήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μπορεί να αλλάξει. Αν υπήρχε μια γενική νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων, ανεξάρτητη από το κατά πόσο γίνονται αντικείμενο ευρεία εμπορία ή όχι, αυτό θα προστάτευε και τα κατοικίδια. Η στρατηγική για την καταπολέμηση των νόσων θα πρέπει να συνδέεται άρεκτα με την στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει ε, δουλειά πάνω σε αυτό. Η διαχείριση των νόσων και η καλή διαβίωση είναι πράγματα άρρηκτα συνδεδεμένα. Η Επιτροπή πάντοτε τα συνδέει, τα έχουν συμπεριληφθεί στις διάφορες εκθέσεις της ΕΦΣΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Όταν λαμβάνεται μία απόφαση για τη διαχείριση ε, Μία νόσου μπορεί να μην λάβει υπόψη πλήρω τον αντίκτυπο που θα έχει στην καλή διαβίωση των ζώων. Αυτό ενίοτε μπορεί να συμβεί ή και το αντίστροφο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα δύο συνδέονται άρρηκτα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το γνωρίζει πολύ καλά. Μιλήσατε για το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Μπορεί κανεί να έχει μια τεράστια γεωργική εκμετάλλευση και να έχει εξαιρετικά καλή διαβίωση των ζώων, εξαρτάται από το σύστημα και το πώς το κάνει δηλαδή ο επιχειρηματίας, ο κτηνοτρόφος. Υπάρχει τάση η επικεφαλής των μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων να χρησιμοποιούν μεθοδολογία η οποία δεν είναι πάντοτε προς όφελος ούτε είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει με, ε, για τα ζώα. Δεν έχω δηλαδή θεμελιώδως καμία ένσταση με το να έχει κανείς μια τεράστια γεωργική κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Μπορεί να την έχει, αλλά πρέπει να υπάρχει νομοθεσία έτσι ώστε και οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις να την ε, ε, πληρούν και να μην μπορούν να ξεφύγουν από αυτήν. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση, σαφέστατα να σας πω ότι διαφορετικά, οι διαφορετικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή δεν πρέπει από τη μία τσέπη να στηρίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι το οποίο από την άλλη δείχνει ότι δεν πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις από άλλο πυλώνα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ελάχιστο είναι να ε, εκπληρεί το σύνολο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας κάτι για να μπορεί να τύχει χρηματοδότησης. Δεν θα πρέπει να ε, χρηματοδοτείτε ή να ανισχύετε ανθρώπους ε, που ασκούν μια εμπορική δραστηριότητα την οποία θα καταδίκαζαν οι περισσότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλους λόγους. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να συνδέεται η να ανισχυετε ανθρωπους που ασκουν μια εμπορικη δραστηριοτητα την οποια θα καταδικαζαν οι περισσοτεροι στην ευρωπαικη ενωση για αλλους λογους ειναι πολυ σημαντικο δηλαδη να συνδεεται η νομοθεσια Δεν λέω κάτι κενό βέβαια υπό το φως του ήλιου. Δεν υπάρχει αυτό. σε κάθε περίπτωση Θέλω να σας πω ότι αναφέρθηκα εσκεμένα στην αηφορία, γιατί όλα αυτά συνδέονται. Ο κόσμος θέλει να δει αηφόρα συστήματα, δηλαδή βιώσιμα, που μπορούν να διατηρηθούν. Θέλουν να δουν την προστασία της φύσης, αυτό θέλει να δει κοινή γνώμη. Την προστασία των ζώων, την καλή τους διαβίωση, χωρίς αντίκτυπο ε, ε, επιβαρυντικό και ευλαπτικό για το περιβάλλον. Άρα, Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα ενιαίο, ολοκληρωμένο. Ε, όταν έχουμε μια αγροτική κτηνιατρική εκμετάλλευση, όταν έχουμε ένα χημικό εργοστάσιο, πρέπει να δούμε τον πλήρη κύκλο, ε, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η αηφορία παντού. Ε, ξέρετε, για τα άγρια ζώα, στο παρελθόν μιλούσαμε για την προστασία της φύσης της Φλωρίδας και της Πανίδας, κυρίως της Πανίδας, χωρίς να μιλήσουμε για καλή διαβίωση. Δεν είναι σωστό να μιλάμε για προστασία της Πανίδας χωρίς μέρημνα για την καλή της διαβίωση. Αν είναι ένα ζήτημα, είναι ζήτημα Πανίδας, ας πούμε αναφερθήκατε στη Φαλαινοθυρία, δεν υπάρχει τρόπος να θυρεύσει κανείς φάλαινες στον οικότοπό τους και είναι διαφορετικό αυτό από ένα ε, δελφίνι ε, που βρίσκεται σε κάποιο ενιδρίο, ακουάριουμ κτλ. Δεν υπάρχει δηλαδή τρόπος να σκοτώσει κανείς μια φάλαινα στον ωκεανό εκεί που διαβιεί ε, φυσικά με καλό τρόπο. Δεν υπάρχει καλή θανάτωση της φάλαινας, δεν υπάρχει τέτοια μεθοδολογία. με τρόπο ανθρώπινο δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα πρέπει αυτά να τα γνωρίζουμε. Και με ρωτήσατε πώς μπορεί να δεχθεί την καλή διαβίωση των ζώων ο ΠΟΕ ως θέμα δημόσιας δεοντολογίας και ηθικής. Πρέπει να σας πω ότι αυτό μπορεί να ισχύσει σε πάρα πολλούς τομείς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αν δεν επιτρέψουμε να έχουμε κότε σε συστοιχίε κλοβών, ε, τότε να μην εισάγουμε αυγά από άλλε χώρε που έχουν γεννηθεί από κότε που σορεύονται σε τέτοιου είδου συστοιχίε κλοβών. Ε, αν δεν επιτρέπουμε εκτροφή ε, ε κρέατος χείρου ε, με αν, παράδεκτες για μας συνθήκες, ε, δεν πρέπει να επιτρέπουμε την εισαγωγή άλλων ε, αντιστοίχων που στις χώρες από τις οποίες εισήχθησαν οι συνθήκες είναι επίσης απαράδεκτες. Όταν μιλούσαμε για το δέρμα της φώκιας, ένα μέρος του επιχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι εμείς δεν παράγουμε ε, δέρμα φώκιας, δεν απαγορεύουμε δηλαδή ε, το εμπόριο αυτό για να προστατεύσουμε τους δικούς μας. Το απαγορεύουμε γιατί θεωρούμε ότι ηθικά δεν είναι σωστό, είναι λάθος και νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα πρέπει να ε, ξαναπροβάλλουμε. Ενδεχομένως είναι δύσκολο να προβληθεί αυτό το επιχείρημα στον ΠΟΕ, αλλά πρέπει να το πράξουμε εάν η νομοθεσία που περνάμε έχει ως πρόθεση να προστατεύσουμε τα ζώα. Νομίζω ότι μπορεί κανεί να έχει μια στέρεα υπόθεση και επιχειρηματολογία στο ΠΟΕ ότι περνάει νομοθεσία όχι για να προστατεύσει τη δική του βιομηχανία, το δικό του κλάδο ω Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για να προστατεύσει την καλή διαβίωση των ζώων. Νομίζω ότι ε, θα έπρεπε να μπορούμε να το κάνουμε και σε παιδεία για τα οποία έχουμε δική μα παραγωγή. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ πολύ για τι ερωτήσει τη πολύ ενδιαφέρουσες, ο πρόεδρο. Και εγώ σα ευχαριστώ. Θα ήθελα να αποδείξω ότι η Προεδρία της Επιτροπής Αναφορών παίρνει στα σοβαρά όλα τα σχόλια που διατυπώνονται στη συνεδρίαση. Κύριε Εκ, αν και να μας είχατε ζητήσει το θάμα του να αλλάξουμε το κόσμο, εμείς θα σας ζητούσαμε τουλάχιστον 24 ώρες να δούμε πώς θα το πράξουμε. Σε κάθε περίπτωση να ακούσουμε ε, την, απο... την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα που θίξατε. Παρακαλώ. Ε, merci, le Président. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την προσπάθεια που κατεβλήθηκε για τη μελέτη αυτή. Να αναφέρω επίσης ότι το 2014 η Επιτροπή είχε ε, ετοιμάσει μια μελέτη για το κόψιμο των ουρών που είχε σημαντικές επιπτώσεις στο έργο της Επιτροπής, διότι έκτοτε διαμορφώθηκε ένα σχέδιο δράσης για το θέμα αυτό, για καλύτερη υλοποίηση της νομοθεσίας. Συνεχίζουμε και είναι ένας από τους βασικούς στόχους της ε, πολιτικής της Επιτροπής. Θέλω επίσης να διευκρινίσω ότι ε, δεν ε, έχω σχόλια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, προσωπικό μου σχόλιο είναι ότι είναι εξαιρετική μελέτη. Ελέγχθησαν αρκετά από ε, τους ευρωβουλευτές για το θέμα αυτό. Εγώ δεν είμαι πολιτικός και δεν μπορώ να μιλήσω για τέτοια θέματα. Αλλά νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει νέα νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν σας λέω τίποτα που δεν ξέρετε. Στα συμπεράσματα τώρα είδαμε αρκετά θέματα και ε, η επιβολή του νόμου είναι ένα από τα θέματα τα οποία και την Επιτροπή την απασχολούν. Όσον αφορά τα επιστημονικά ζητήματα και τη διάδοση των επιστημονικών γνώσεων, συμφωνεί απολύτως η Επιτροπή με τα συμπεράσματα της μελέτης. και μετά την έγκριση του κανονισμού για τους επισήμους ελέγχους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δημιουργήσει κάποια κέντρα αναφοράς για την ορθή διαβίωση των ζώων περίπου ένα έτος μετά την ε, δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα. Είναι λοιπόν ε, κάτι το οποίο ήδη προχωρεί στην Επιτροπή. Και να προσθέσω και κάτι ακόμη. Όπως είπαμε, δεν είναι καθόλου πιθανόν να προκύψει νέα νομοθεσία, αλλά ο Επίτροπος έχει ήδη ανακοινώσει ότι από τα τέλη Ιανουαρίου έχουμε μια πλατφόρμα για την ορθή διαβίωση των ζώων και 6 Ιουνίου θα γίνει μια πρώτη συνεδρίαση. Εξαρτάται λοιπόν από τη βούληση των εμπλεκομένων, αλλά όλοι έχουν να παίξουν ένα ρόλο για αυτό το θέμα. Η ορθή διαβίωση των ζώων μας αφορά όλους, δεν είναι μόνο το έργο των θεσμικών οργάνων, αλλά είναι και η προσπάθεια του καθενός από εμά. Και έχοντας δουλέψει πάνω σε αυτό το θέμα πάνω από 15 χρόνια, βλέπω σήμερα ότι είναι όριμο το θέμα ε, και για τις οργανώσεις προστασίας των ζώων και για τους επιστήμονες και για τις επιχειρήσεις. Όλοι προσπαθούν να συνεργαστούν για κοινά σχέδια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χάζενκαμ. Αλλά να είστε σύντομοι, παρακαλώ. Άκουσα τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μα είπε ότι δεν έχει συγκεκριμένη εντολή να μιλήσει εκ μέρου τη Επιτροπή για αυτή τη σημαντική έκθεση. Προτείνω η Επιτροπή Αναφορών να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία επίσημη αντίδραση για την έκθεση αυτή, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα για να το αφήσουμε έτσι και απλώς να μας λέει η Επιτροπή ότι δεν έχει εντολή να απαντήσει. Πρόεδρος, συμφωνώ. Να προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, λοιπόν. Ο κύριος Εκ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε άλλη μια φορά το λόγο. Δεν περιμένω θαύματα από την Επιτροπή Αναφορών. Κάθε άλλο. Αντιθέτως, χαιρετίζω το ότι είναι τόσο αποφασιστική η Επιτροπή Αναφορών και ασχολείται με αυτό το θέμα. Αλλά είναι και καθήκον της Επιτροπής Αναφορών. να συγκεντρώνουμε ένα τέτοιο όγκο αναφορών από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να δείξουμε ότι αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα της προστασίας των ζώων και της ορθής διαβίωσης των ζώων για τον λαό της Ευρώπης. Και προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε συνηθίσει στο μπλα μπλα της Επιτροπής. Θέλουμε να έχουμε κάτι ξεκάθαρο, κάτι ουσιαστικό. Ε, δεν θέλουμε ομιλίες επί ομιλιών, όχι λόγια, έργα. Ευχαριστώ. Νομίζω τώρα, κυρίες και κύριοι, λέει ο θα πρέπει να ασχοληθούμε με κάποιες αναφορές. Έχουμε την ε, αναφορά της κυρίας Ανίκ Πιλάχ, υπαριθμών 820 του 2015, δεν είναι παρούσα η αναφέρουσα, αφορά την απαγόρευση παγίδων με κόλλα για ε, τα τροκτικά. Θα ήθελα να ζήσω τον κύριο Σιπριάνη να λάβει το λόγο για την αναφορά αυτή. Καλημέρα σας. για να σας περιγράψω το πλαίσιο της αναφοράς αυτής. Πρόκειται για μία αναφορά που ζητάει απαγόρευση συγκεκριμένου τύπου παγίδας, παγίδας κόλλας που χρησιμοποιείται για τη σύλληψη τροκτικών. Πρόκειται για μικρές πλαστικές πλάκες με μία στρώση κόλλας. Σε κάποια κράτη-μέλη στο εμπόριο, ενώ σε άλλα κράτη-μέλη απαγορεύονται για λόγους ε, καλή διαβίωση των ζώων. Έχουμε λοιπόν διαφοροποιημένη κατάσταση εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το πρόβλημα των παγίδων αυτών είναι ότι είναι πολύ αποτελεσματικές ε, για τη σύλληψη των τροχτικών και χρησιμοποιούνται ευρέως σε κάποιες χώρες. θεωρείται απάνθρωπη η μέθοδος αυτή, διότι τα ζώα δεν σκοτώνονται αμέσως. Μπορούν έτσι να έχουν έναν πολύ αργό και βασανιστικό θάνατο. Σίγουρα λοιπόν πρόκειται για θέμα καλής διαβίωσης των ζώων. Ε, τα ποντίκια όμως και οι αρουραίοι είναι άγρια ζώα, δεν είναι κατοικίδια και δεν καλύπτονται από καμία νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε, για παράδειγμα, ε, τις ε, οδηγίες για τα πτηνά ή για τους ε, οικότοπους. Δεν πρόκειται για νομοθεσία για την προστασία των ζώων, είναι νομοθεσία για την προστασία της βιοπικιλότητας. Σαφώς ε, λοιπόν τα τροκτικά βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογή οποιασδήποτε ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσον αφορά τη διατήρηση ε, ή την ε, καλή διαβίωση, την προστασία των ζώων. Η αναφέρουσα επίσης αναφέρει ότι σε κάποιες περιπτώσεις συλλαμβάνονται εκεί και άλλα είδη προστατευμένα, αλλά είναι τόσο ελάχιστες ε, οι περιπτώσεις αυτές που σίγουρα δεν μπορούμε ε, να χρησιμοποιήσουμε την νομοθεσία για την διατήρηση των ειδών ε, για να απαγορεύσουμε αυτές τις παγίδες. Είναι λοιπόν καθαρά θέμα καλής διαβίωσης των ζώων για τη σύλληψη ζώων μη κατοικιδίων. Δεν υπάρχει νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να καλύπτει το θέμα αυτό. Είναι λοιπόν θέμα εκτός πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας μας και παραμένει θέμα εθνικής νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτον, να δώσω το λόγο στους συναδέρφους, θα ήθελα να ρωτήσω τον, ε, τον κύριο καθηγητή ποια είναι η δική σας θέση ως εμπειρογνώμονα για την ε, αναφορά αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επί αρκετά χρόνια εκπροσωπούσα την Ευρωπαϊκή Ένωση στις συζητήσεις με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η ε, Κίνα, πριν 10-15 χρόνια. Και όσον αφορά τις παγίδες και υπάρχει κάποια ε, νομοθεσία για παγίδες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι παγίδων που δεν επιτρέπονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω λοιπόν πείρα στο θέμα αυτό. Σίγουρα φαίνεται σαν ε, να είναι ανομαλία το να επιτρέπουμε ε, παγίδες που είναι εξίσου κακές με παγίδες απαγορευμένες είναι καταρχάς πολύ δύσκολο να, καθορίσει, να ρυθμίσει κανείς ε, την ε, παγίδα για να μην ε, ε, συλλαμβάνονται και προστατευμένα είδη. Για παράδειγμα, μπορεί να συλληθούν τυφλοπόντικες, πτηνά, μερικές φορές κατοικίδια ζώα. Αλλά βέβαια θα πρέπει να πρόκειται για πολύ μικρά κατοικίδια ζώα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι πρόκειται για μέθοδο σύλληψης ε, που δεν κάνει διακρίσεις. Το δεύτερο θέμα είναι ότι όταν ε, συλλαμβάνονται τα ζώα αυτά, τα ζώα αυτά υποφέρουν εξίσου με άλλα ε, είδη τα οποία προστατεύουμε. Τα ποντίκια έχουν συστήματα πόνου και τρόμου είναι λοιπόν πολύ σημαντική η ε, ανταπόκριση των συστημάτων αυτών όταν συλλαμβάνεται ένα ζώο σε μια τέτοια παγίδα. Τι γίνεται λοιπόν, ε, εάν είναι χαμηλή θερμοκρασία, τα ζώα αυτά πεθαίνουν από ε, το κρύο. Σε περιπτώσεις που παραμένουν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πεθαίνουν από την πείνα. Είναι λοιπόν παγίδες με πολύ αρνητικές συνέπειες για την καλή διαβίωση των ζώων αυτών. Δεν υπάρχει λοιπόν ε, κανένα καλό επιχείρημα για τη χρήση τους, εκτός του ότι λειτουργούν καλά. Θα πρέπει να προστατεύουμε τα ζώα, των οποίων τον αριθμό θέλουμε να ελέγξουμε. Το ότι πρόκειται για ε, βλαβερά ζώα δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της διαβίωσής τους. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικά θέματα καλής διαβίωσης, προστασίας των ζώων. Ε, συχνά συλλαμβάνονται ζώα τα οποία δεν θέλουμε να σκοτώσουμε και σίγουρα δεν πρόκειται για ανθρώπινο τρόπο θανάτωσης των ζώων αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Πέτερ Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να τονίσω μια άλλη πτυχή που συνδέεται και με την μελέτη που ακούσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα αναφερόμαστε στην εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς. Ε, το... Τέτοια θέματα λοιπόν έχουν προκύψει αρκετά αργά στο θεματολόγιο, κυρίως ε, ασχολούμασταν με εμπορικά θέματα. Σε πολλά κράτη-μέλη λοιπόν δεν επιτρέπονται αυτές οι παγίδες κόλαση, σε άλλα κράτη-μέλη επιτρέπονται. Ε, εγώ θα θεωρούσα ότι είναι θέμα εσωτερικής αγοράς. Είναι αφελές να πιστεύουμε ότι αν επιτρέπονται Τρέπεται η πώληση της παγίδας αυτής σε ένα κράτος μέλος, ε, μπορώ να την αγοράσω και να τη χρησιμοποιήσω αλλού. Θα πρέπει λοιπόν τα άλλα κράτη-μέλη να σκεφτούν ότι δεν μπορούν να εφαρμόσουν την απαγόρευσή τους ε, επειδή μπορεί να αγοράσει κανείς αλλού την παγίδα αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να Προτείνω να κλείσουμε την αναφορά αυτή ναι, να ε, παρακολουθήσουμε όμως ε, την κατάσταση στην εσωτερική αγορά. Το να επιτρέπεται η παγίδα αυτή σε ένα κράτος μέλος και να απαγορεύεται σε άλλο ε, δεν έχει νόημα, διότι υπάρχει η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να κλείσουμε την αναφορά αυτή και να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για θέμα εσωτερική αγορά. Χωρί βέβαια να αμφισβητώ αυτά που είπατε εσεί, πολύ σωστά ήταν, αλλά έχουμε ε, διαφορετικέ ε, νομοθεσίε εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Η κυρία Εύη. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως. είναι και θέμα εσωτερικής αγοράς. Εκτός από τη βοήθεια που πρέπει να δώσουμε για την καλή διαβίωση των ζώων. Πράγματι υπάρχουν διαφορετικές νομοθεσίες, πράγματι είναι κατακαιρματισμένη η αγορά. Αναρωτιέμαι όμως, αφού υπάρχουν εναλλακτικέ, πολύ καλύτερες, που δεν προκαλούν ούτε τη θανάτωση ούτε την οδύνη του ζώου. Γιατί δεν προσπαθούμε και σε αυτό το πλαίσιο να προωθήσουμε αυτές τις εναλλακτικέ. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται εδώ λόγος για ζώα που δημιουργούν ε, προβλήματα δημόσιας υγείας και υγιεινής. Ε, άρα θα πρέπει να έλεγχε το πληθυσμό τους αφέστατα. Αυτό είναι κατανοητό. να απαγορεύσουμε αυτές τις παγίδες και να προωθώσουμε διαφορετικές λύσεις στα διάφορα κράτη-μέλη, να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό της αγοράς και να ενισχύσουμε ε, την καλή διαβίωση των ζώων. Να κρατηθεί ανοιχτή αναφορά, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ λέω να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά όπως είπε ο καθηγητής γιατί είναι ένας βασανιστικός τρόπος θανάτου. Το, να έχουμε μια παγίδα με κόλλα πάνω στην οποία ε, συλλαμβάνεται ένα ζώο δεν έχει καμία σχέση με τη σύγχρονη Ευρώπη και τις σύγχρονες πρακτικές. Και όπως είπε και ο Πίτα Γιάχ, θέλουμε να έχουμε ένα, μια εναρμόνιση στην Ευρώπη, να υπάρχει ένας χώρος όπου υπάρχουν, ε, υπάρχει ίση βάση, έχουμε τις ίδιες βασικές αρχές και να υπάρχουν κάποιες ηθικές αξίες οι οποίες θα λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα κράτη-μέλη. Και εγώ λοιπόν συμφωνώ να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Παρακαλώ, κυρία Άουκεν. Έχω ασχοληθεί και εγώ πολύ με την ορθή διαβίωση των ζώων και κατά την προετοιμασία μου έκανε εντύπωση που επιμένει η Επιτροπή ότι δεν είναι αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα έχουμε σχετική νομοθεσία Είχαμε κάνει αρκετές συνεδριάσεις ε, για τους χείρου, για το κόψιμο της ουράς και για τις συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να γίνεται και για τη βιομηχανική εκτροφή. Μπορεί να μην είναι το πλέον σημαντικό, αλλά σαφώς ε, εντάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και μου κάνει εντύπωση και είναι και ανησυχητικό που η Επίτροπη δεν κάνει τίποτα επ' αυτού. σχετικά με τα τροκτικά στη Δανία. Είχα ασχοληθεί με τις ε, δοκιμές που γίνονται στα ζώα και ήμασταν πάρα πολύ αυστηροί για την μεταχείριση των ζώων συμπεριλαμβανομένων των αρουραίων. Δεν ε, επιτρέπεται να προκαλούμε πόνο ακόμη και αν πρόκειται για έναν ε, αντιπαθητικό αρουραίο. Ακολουθούσαμε και κάποιους κανόνες του ΩΣΑ στη Δανία αλλά και στην κοινωτική νομοθεσία πρέπει να έχουμε κάτι. Δεν καταλαβαίνω γιατί λέει η Επιτροπή ότι δεν έχει καμιά δουλειά με κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Προτείνω την εξή λύση. Ας κρατήσουμε καταρχήν ανοιχτή την αναφορά, διότι πρόκειται για πραγματικό πρόβλημα. Δεύτερον, θα στείλουμε δύο επιστολές. Μία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μία δεύτερη προς την Επιτροπή ΙΜΚΟ, όπου θα τους ενημερώνουμε για τις σημερινέ μας συζητήσει. για το ότι απαιτείται, κατά τη γνώμη μας, εναρμόνιση της νομοθεσίας σε αυτό το θέμα και θα δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτό το θέμα με βάση τα αποτελέσματα των επιστολών μας. Δεύτερον, το επόμενο θέμα είναι η τελετουργική σφαγή. Αναφορές που υποβάλλονται από πολίτες στην Πολωνία, Γαλλία και Γερμανία. Δεν είναι παρόντες οι αναφέροντες. Θέλω να ζητήσω από τον Τένι Σίμωνιν από την Γενική Διεύθυνση Σαντέ να λάβει το λόγο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συνοψίσω λίγο το θέμα. Οι αναφορές ζητούν ε, την κατάργηση της θανάτωσης χωρίς αναισθητοποίηση στο πλαίσιο τελετουργικών σφαγών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απαντήσει πολλές φορές δίνοντας την ίδια απάντηση, δηλαδή δεν προτίθεται η Επιτροπή να τροποποιήσει τα εφιστάμενα κείμενα, διότι οι διατάξεις αυτές που επιτρέπουν την τελετουργική σφαγή πλαισιώνονται με κάποια τεχνικά μέτρα και το πιο σημαντικό είναι ότι επιτρέπουν την ισορροπία μεταξύ αφενός μεν της υποχρέωσης για ορθή διαβίωση των ζώων, αφετέρου δε ε, της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στην οποία, την οποία έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την εγγύηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων. Ε, επιτρέπει λοιπόν μια ισορροπία μεταξύ των δύο. Τώρα πρέπει να τονίσουμε ότι το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει λεπτομερείς διατάξεις για την εφαρμογή της τελετουργικής σφαγής στα σφαγεία, διότι σε μεγάλο βαθμό εξατάται από την εκτίμηση των κρατών μελών, καθώς οι συνθήκες διαφέρουν σε κάθε χώρα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε καθηγητά, μπορείτε να μας πείτε τη γνώμη σας. Ευχαριστώ. Όπως γνωρίζει πολύ καλά ο Ντενή Σίμωνα, υπάρχουν πάρα πολύ καλά στοιχεία ε, σχετικά με την τελετουργική σφαγή και από τη στιγμή που ε, κόβεται ο λαιμός, ε, η, επιβίωση, η, η διαβίωση των ζώων ε, δεν είναι καλή. Εξαρτάται από το είδος του ζώου. Μπορεί να είναι δύο λεπτά στα βοηδή και στα κοτόπουλα και λίγο λιγότερο στα πρόβατα. Είναι διάστημα κατά το οποίο υποφέρουν πολύ τα ζώα. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι αν γίνει η τομή και αναισθητοποιηθεί το ζώο κατά την ίδια στιγμή, το, το ζώο χάνει το αίμα του. Η αφέμαξη είναι το θέμα για τα θρησκευτικά ζητήματα. Η αφέμαξη γίνεται ε, ε, ακόμη και αν αναισθητοποιηθεί το ζώο. Δηλαδή, αν το αναισθητοποιήσουμε, δεν σταματάμε την αιμορραγία. αλλά εφόσον το ζώο χάνει το αίμα του, επιτυχάνεται ο σκοπό τη τελετουργική φαγή. Για πολλού, ιδίω για τι μουσουλμανικές κοινότητε, θα πρέπει να φροντίσουμε να πισθούν, να γίνεται η τομή του λαιμού μαζί με την αναισθητοποίηση. Πολλέ φαγέ χαλάλ γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Αναισθητοποίηση και τομή ε, ε, στο λαιμό κατά, τον ίδιο, κατά την ίδια στιγμή. Κάποιες μουσουλμανικές κοινότητες ε, λοιπόν ε, έχουν δεχθεί την ε, πίεση της κοινή γνώμης γιατί η κοινή γνώμη πιστεύει ότι είναι απάνθρωπο να σκοτώνουμε το ζώο χωρίς να το έχουμε αναισθητοποιήσει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νομοθεσία για την διαβίωση των ζώων είχε επιβάλλει αναισθητοποίηση πριν από τη σφαγή ήταν από τα πρώτα πράγματα που είχαμε κάνει και τώρα φαίνεται ε, ε πραγματικά φρικτό να υπάρχουν ζώα τα οποία θανατώνονται χωρίς αναστητοποίηση. Καλό θα ήταν λοιπόν να πείσουμε τις θρησκευτικέ κοινότητες ότι μπορούν να κάνουν αυτές τις αλλαγές στον τρόπο τελετουργικές σφαγές και πρέπει να τονίσουμε ότι σε ορισμένε χώρες ήδη γίνεται. Από, από επιστημονικής πλευράς είναι σίγουρο ότι το ζώο υποφέρει και μπορεί να υποφέρει για μέχρι δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Άουκεν. Εγώ ήμουν στο Κοινοβούλιο στη Δανία επί 20 χρόνια και αυτό ήταν ένα θέμα που το συζητούσαμε ξανά και ξανά. Στη Δανία οι μουσουλμανικές κοινότητες δέχθηκαν την αναισθητοποίηση. Εδώ και χρόνια το έχουν δεχτεί, ούτω ώστε πριν τη σφαγή των ζώων να υπάρχει η αναισθητοποίηση. Αποδείχθηκε ότι υπέφεραν τα ζώα. Το πρόβλημα εδώ είναι ποια θρησκευτική κοινότητα έχει τέτοιες τελετουργικές φαγές. οι μουσουλμάνοι έχουν δείξει προθυμία να προσαρμοστούν. Δεν ξέρω μήπως άλλες ε, θρησκευτικές κοινότητες δεν το δέχονται. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιμείνουμε ότι πρόκειται για επιστημονικά δεδομένα που αποδεικνύουν ότι το ζώο υποφέρει. Δεν, έχουμε, δεν έχει καμία σχέση με την ανεξιθρησκεία. Ε, Όλοι συμφωνούμε με την ελεύθερη άσκηση της θρησκείας. Υπάρχει ελευθερία άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων, αλλά υπάρχουν ε, και υπάρχουν διάφορα κρεοπολία που πουλάνε ε, κρέας με βάση διαφορετικές συνήθειες, χαλάλ ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά εκτός από την τεχνική χαλάλ υπάρχει και η τεχνική σέκνιν που δεν χρησιμοποιούν αναισθητοποίηση και νομίζω ότι αυτό περισσότερο αποτελεί πρόβλημα. Εγώ είμαι θεολόγος και έχω διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη και ε, τις τελετουργικές φαγές έχω διαβάσει ότι πρόκειται για τεχνικές που ζητούν ένα ακέραιο ζώο. Δεν επιτρέπεται λοιπόν η αναισθητοποίηση, αλλά στην Παλαιά Διαθήκη δεν λέει πουθενά ότι πρέπει να υποφέρει το ζώο. Είναι θεολογικά επιχειρήματα αυτά τα οποία αναφέρω τώρα. Ξέρετε μήπως σε ποιες χώρες έχει σταματήσει αυτή η θανάτωση χωρίς καμία μορφή αναισθητοποίησης. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι η ώρα να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με αυτές τις αναφορές. Ο κύριος Εκ. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά την ε, σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση, θα πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο θα δούμε όλο και περισσότερο στο μέλλον στην Ευρώπη. Θα δούμε Μάλλον έχει αυξηθεί η προσέλευση ε, πολιτών από άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είδαμε αυτό ως αποτέλεσμα του πολέμου ε, στη Μέση Ανατολή και πρόκειται μόνο για την κορυφή του παγόβουνου ε, σε σχέση με όλους όσους θα καταφτάσουν λόγω της αλλαγής του κλίματος, διότι θα έρθουν μετανάστες πείνας πια και θα δούμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό μουσουλμάνων στην ε, Ευρώπη που θα θέλουν κρέας χαλάλ. Και τίθεται το θέμα αν θα πρέπει να το δεχτούμε ή όχι. Ο καθηγητής Μπρούμ το ανέφερε αυτό και εγώ έχω δει πολλές ταινίες για την τελετουργική σφαγή. Ε, είναι ε, απάνθρωπος τρόπος σφαγής, συχνά και δεν τηρούνται οι κανόνες της υγιεινής. Και η διαδικασία θανάτου διαρκεί μερικές φορές μέχρι, σε, μέχρι και ακόμα 10 λεπτά. Ε, κόβουν την καροτίδα του ζώου και το ζώο ε, προσπαθεί σε κάποιες περιπτώσεις να διαφύγει. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε ε, το θέμα του βασανισμού των ζώων, από την άλλη έχουμε το θέμα της ε, ανεξιθρησκεία. Αλλά όσον αφορά την ανεξιθρησκεία, την ελευθερία μάλλον άσκησης ε, της θρησκείας, οι μουσουλμάνοι πιστεύουν στην Σαρία που είναι ένας πολύ αυστηρός κώδικας κανόνων για τους πιστούς. Στην Ευρώπη όμως απαγορεύεται αυτό, λέμε, απαγορεύεται το μαστίγωμα των γυναικών κλπ. Ε, στα ζώα όμως τα επιτρέπουμε. Βλέπουμε και πάλι αυτήν ε, ε, την διάκριση, πώς λαμβάνουμε διαφορετικές αποφάσεις όταν αφορούν τους ανθρώπους ή όταν αφορούν τα ζώα. Στα ταξίδια που έχω κάνει, το έχω δει. Ε, εκατομμύρια ανθρώπων υποφέρουν όμως άλλωστε όταν ε, βλέπουν ε, πώς γίνονται οι σφαγές με τρόπο χαλάλ. Ε, άλλωστε, εγώ τόσα χρόνια ζω, είμαι απόλυτα υγιής, χωρίς ε, κρέας. ούτε τους μουσουλμάνους θα τους βλάψει αυτό. Παρακαλώ λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή. Όχι, όχι. Πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε το θέμα αυτό μέχρι να φτάσουμε σε καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πέτερ Γιάρ. Ευχαριστώ. Συμφωνούμε εδώ στην αίθουσα ότι πρόκειται και για θέμα εξωτερικής πολιτικής και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν αφορά μόνο τους μουσουλμάνους, αφορά και τους Εβραίους. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο το θέμα αυτό και ο καθηγητής ίσως είπε τη σωστή λέξη. Είτε το πες και εμένα είτε όχι. Θα πρέπει να βοηθήσουμε, να πείσουμε και όσον αφορά τη θρησκεία. Δέχτηκα στο γραφείο μου φοιτητή που μου ζήτησε η υποστήριξη της Ευρώπης για το θέμα αυτό. Πρέπει να συζητήσουμε το θέμα. Ούτε θα βρούμε γρήγορα κάποια λύση. Αλλά μου φαίνεται υπερβολικά εύκολη λύση απλά να κλείσουμε την ε, αναφορά. Χρειάζεται να γίνει η σχετική συζήτηση. Πρόκειται για θέματα Ε, βαθύτατα θρησκευτικά, τα πράγματα κινούνται πολύ αργά. Εγώ όμως ε, θέλω να πιστεύω ότι ε, κάποια στιγμή μετακινούνται και οι θέσεις. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσουμε τη συζήτηση και να λύσουμε το πρόβλημα από τη μία της προστασίας των ζώων και από την άλλη της ελευθερίας στην θρησκεία. Άλλωστε είναι πολιτικό το θέμα, μην αυταπατώμεθα. Köszönöm oh, Ερωτήσεις έχετε. Ναι. Όλοι οι μουσουλμάνοι στη Δανία έχουν καταργήσει τη σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση, χρησιμοποιούν το πιστόλι αναισθητοποίησης. Όμως, σε πόσες χώρες οι εβραϊκές κοινωνίες δέχτηκαν να σταματήσουν το σέκνινγκ, ε, την τεχνική αντίστοιχη χωρίς αναισθησία. Μήπως το ξέρετε, ο κύριος Μπρούμ. Δεν το ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Νομίζω ότι οι μουσουλμανικές κοινωνίες απάντησαν λέγοντας ότι θα αλλάξουμε και σε γενικές γραμμές νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες δεν άλλαξαν. Ίσως κάποιες έχουν αλλάξει και να μην το ξέρω. Εγώ δεν έχω τέτοιες πληροφορίες. Δεν ξέρω να έχει αλλάξει κάποια από αυτές. Όμως πρέπει να σας πω ότι παρέστην σε μια σύσκεψη στο Λονδίνο και εκεί υπήρχαν εκπρόσωποι και εβραϊκών και μουσουλμανικών κοινοτήτων και σίγουρα εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να λυθεί το πρόβλημα και στις δύο κοινότητες. Και γίνεται συζήτηση για τις συνέπειες της διαδικασίας αναισθητοποίησης και ποια επίπτωση θα έχει αυτό στο κρέας και νομίζω ότι τώρα οι εβραϊκές κοινότητες δέχονται όλο και περισσότερο ενδεχομένως ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι αγνό στην αναισθητοποίηση και ότι η αναισθητοποίηση δεν το προκαλεί, δεν προκαλεί ε, το κρέας, δεν κάνει το κρέας να ε, μην γίνεται, να μην παραμένει αγνό. Βεβαίως μέρος, μέρη ε, των ε, ζώων αυτών πολλούνται και σε ανθρώπους που δεν ανήκουν στην εβραϊκή κοινότητα. Άρα το προϊόν αυτό μπαίνει στην αγορά την γενικότερη χωρίς σήμαση. Και έτσι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να φάνε ένα ζώο που δεν αναισθητοποιήθηκε πριν σφαγιαστεί, τελικά καταλήγουν να τρώνε ζώο που δεν αναισθητοποιήθηκε ε, πριν σφαγιαστεί, γιατί δεν υπάρχει επαρκή σήμανση, ε, γιατί δεν μπορεί να πεταχθεί αυτό το κρέας και όσοι το σφαγιάζουν με την, ε, τον τρόπο αυτό, τελικά τα υπόλοιπα όσα δεν καταλώνονται τα θέτουν σε ευρεία εμπορία και δεν θα πρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πει ότι ε, στη Δανία πολλούμε πάρα πολύ κρέας χαλάλ και όλα έχουν αναισθητοποιηθεί και δεν ισχύει η θρησκευτική διάσταση. Ε, το μας ενδιαφέρει το να μην υποφέρει το ζώο. Όχι ε, τι προσευχή διαβάζεται πριν σφαγεστεί βάσει της μεθόδου χαλάλης έκνικ. Το θέμα της αναισθητοποίησης λοιπόν επιβλήθηκε και η εβραϊκή κοινωνία μας έλεγε ότι ε, με το χτύπημα του πιστολιού στο κεφάλι πλήττεται το ζώο το οποίο είναι χτύπημα επιστολού για αναισθητοποίηση. Θεωρώ ότι αυτή η υπερχηματολογία είναι αρκετά ε, θεμελιακή, φονταμενταλιστική ενδεχομένως. Να είμαστε προσεκτικοί, να μην δακτυλοδείχνουμε τους μουσουλμάνους, γιατί έχουν συμμορφωθεί εδώ και δεκαετίες και κινούνται, δραστηριοποιούνται εδώ και πολύ καιρό. Ο πρόεδρος. Πράγματι, Από τη στιγμή που δεν παρίστανται οι ραβίνοι και οι, οι, μάμιδες, η, στη συζήτηση πρέπει να την κάνουμε εμείς. Δεν το θεωρώ ότι είναι ένα θέμα θρησκευτικής ελευθερίας. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Νομίζω ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός υπάρχει, είναι σημαντικός και ζητούμε από όλους να σέβονται ε, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Το ίδιο ισχύει και με τη θανατική ποινή. Στην Ευρώπη δεν μπορεί να είναι αποδεκτή η θανατική ποινή. Η Ευρώπη έχει κάνει διάφορα βήματα προς τα αυτό, που θα μπορούσε να κάνει και περισσότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, δεν μπορούμε να δεχθούμε να επανεισαχθεί η θανατική ποινή γιατί αυτό δεν είναι μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού, δεν ταιριάζει με το αξιακό μας σύστημα. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο ισχύει και σε αυτή την περίπτωση και δεν υπάρχει σχέση με θρησκευτική ελευθερία. Αν κλείσουμε αυτή την αναφορά τώρα δεν ασκούμε πίεση ούτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε στις θρησκευτικές κοινότητες. Ο κύριος καθηγητής είπε κάτι το πολύ σημαντικό και είπε ότι το έχω συζητήσει και με επικεφαλής των Ευρωπαϊκ... εβραϊκών κοινοτήτων και με επικεφαλής των μουσουλμανικών κοινοτήτων και μου είπαν ότι ενδιαφέρονται να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα. Άρα αυτές οι κοινότητες ενδιαφέρονται να λύσουν αυτό το πρόβλημα με πιο πολιτισμένο τρόπο. Άρα αν κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή, είναι ο τρόπος μας να ασκήσουμε μια κάποια πίεση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να συντάξουμε μια επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημερώνοντάς τη ότι κρατούμε την αναφορά ανοιχτή και ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει το κατά πόσο μπορούμε να περάσουμε σε υψηλότερα νομοθετικά επίπεδα. Εάν συμφωνείτε, προχωράμε στην αναφορά 1542 του 2010 και την προστασία ε, της Αρκούδας, της καφέ Αρκούδας, Φρανσουά Arcangeli, ο αναφέρον και έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη σύνοψη της κατάστασης της καφέ Αρκούδα στα Γαλλικά Πυρηναία. Θέλω να διευκρινίσω ότι είναι ένα είδος το οποίο αποτελεί προτεραιότητα σε κοινωτικό επίπεδο και απαιτείται προστασία περιοχών και ζωνών ε, ειδική διατήρησης. Είναι ζώνες που μπαίνουν στο Natura 2000 βάσει της οδηγίας για τους βιότοπους και οικότοπους, οδηγίας Habitat. Είναι ένα καθεστώς αυστηρής προστασίας ε, για να μην διαταραχθεί το είδος. Ε, μελετήσαμε επισταμένως τις εξελίξεις το πώς εξελίσσεται η καφέ αρκούδα στα Πυρηναία τα τελευταία χρόνια. Επανησύχθηκαν ε, κάποια ζώα από τη Σλοβενία και απελευθερώθηκαν στα γαλλικά Πυρηναία για να ζήσουν ελεύθερα. Ο πληθυσμός τους άρχισε λοιπόν να αυξάνεται. Η επανεισαγωγή της καφέ αρκούδας έγινε στη δεκαετία του 90, από το 96 μέχρι το 2006 και έχει βελτιωθεί η ποσοτική εκπροσώπηση του είδους στο ε, ε, στον κεντρινό ορεινό όγκο των Πυρηναίων, ενώ στα δυτικά έχουμε μόνο δύο αρσενικές καφέ αρκούδες, άρα το είδος απειλείται με εξαφάνιση, έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Άρα, ε, στον κεντρινό ορεινό όγκο έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά όχι αλλού. Τώρα το θέμα είναι η ποιότητα. Επειδή δεν υπάρχει μεγάλη γενετική μίξη στην αναπαραγωγή της καφέ αρκούδας, θεωρούμε ότι οι πληθυσμοί θα, αρχίσουν να αποδυναμώνονται σε βάθος χρόνου. Και σύμφωνα με τις πρόσφατες επιστημονικές μελέτες θα πρέπει να επανεισάγουμε στα πυρηναία θηλυκά ζώα από τη Σλοβενία για να υπάρξει γονιδιακό ανακάτεμα που θα ενισχύσει ε, το είδος αυτό για να γίνει πρέπει να ληφθεί αντίστοιχη πολιτική απόφαση. Τώρα το 2012 ξεκίνησε μια διαδικασία επιπαραβάση που είχε κυρίως να κάνει με τους κανόνες ε, ε, για θύρευσης και υπ' αυτή την έννοια Έκτοτε οι γαλλικές αρχές βελτίωσαν το καθεστώς ε, του κυνηγιού στα Πυρηναία για την προστασία της καφέ Αρκούδας και λύθηκε το πρόβλημα της ε, διατάραξης. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να πάρουν οι γαλλικές αρχές για να παρεμποδίσουν, παρεμποδίσουν περαιτέρω επιδίνωση της κατάστασης του είδους της καφέ αρκούδα στα Πυρηναία, Χρειάστηκε να περάσει κάποιος χρόνος μέχρι ότου η Γαλλία να μας ενημερώσει για τα μέτρα που προτίθεται να υιοθετήσει. Υιοθέτησε ένα σχέδιο διαχείρισης του είδους που ολοκληρώθηκε το 2009. Οι γαλλικές αρχές επανειλημμένως ανακοίνωσαν ότι επρόκειτο να υιοθετήσουν μέτρα για τη συνέχιση και αντικατάσταση αυτού του σχεδίου διαχείρισης του πληθυσμού της καφέ Αρκούδας στα Πυρηναία σε συνένεση και διαβούλευση με τις τοπικές περιφερειακές αρχές και με τον τοπικό πληθυσμό και πρόσφατα μας ανακοίνωσε η Γαλλία ότι ένα προσχέδιο σχεδίου δράσης έχει εγκριθεί, έχει μπει στη δημόσια διαβούλευση και ότι τώρα ε, το μπαλάκι βρίσκεται στην πλευρά των γαλλικών αρχών οι οποίες θα λάβουν υπόψη τους ε, τις γνώμες των διαφόρων έτσι όπως θα κατατεθούν στη δημόσια διαβούλευση και των συμβουλευτικών αρχών και θα προχωρήσουμε μετά στην έγκριση του τροποποιημένου σχεδίου. Η Επιτροπή περιμένει με ανυπομονησία επιτέλους την έγκριση αυτού του σχεδίου διαχείρισης του πληθυσμού της καφέ Αρκούδας για να μπορέσει να αποφανθεί το, για το κατά πόσο τα μέτρα για τη διατήρηση του πληθυσμού είναι τα αναγκαία και τα κατάλληλα για να ε, μπορέσει να επιβιώσει η καφέ Αρκούδα σε πιο ευνοϊκές συνθήκες. Περιμένουμε λοιπόν να λάβουμε αυτό το σχέδιο διαχείρισης για να δούμε κατά πόσο θα κλείσουμε τη διαδικασία επί παραβάση ή θα την επανεκκινήσουμε επί τη βάση του άρθρου 6,1 της οδηγίας Habitat για ε, λόγους έλλειψης υιοθέτηση απαραίτητων μέτρων για τη διατήρηση του είδους της καφέ αρκούδα στα Πυρηναία. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, σας δίνω πάλι το λόγο. Ποιος είναι, ποια είναι η γνώμη σας ως εμπειρογνώμων. Δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Καταρχάς, οι αρκούδες μετακινούνται αρκετά και είμαι βέβαιος ότι οι εκπρόσωποι της Κομισιόν το γνωρίζουν αυτό. Αυτό το γεγονός όμως δυσκολεύει τη διαχείρισή τους, διότι θα πρέπει να προστατεύονται σε μια ευρύτερη περιοχή. Και η άλλη παρατήρηση είναι ότι αν μετακινούνται, για να μετακινούνται από ένα μέρος σε άλλο, χρειάζονται ασφαλείς περιοχές. Δηλαδή, χρειάζονται λωρίδε δασών στι οποίε να μπορούν να μετακινούνται ώστε να μην βγαίνουν σε μέρη ανοιχτά. Μέρο λοιπόν τη διαχείριση είναι τρόποι να μετακινούνται από το ένα μέρο στο άλλο ε, και επίση ε, πρέπει να ε, εμποδίζουμε του ανθρώπου να τι βλάπτουν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πέτεριά, παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε πολύ σωστά ότι θα εξετάσει το, μέτρο, το σχέδιο διαχείρισης ε, των γαλλικών αρχών και θα αποφασίσει αν αυτό αρκεί. Υποθέτω ότι θα το ξαναδούμε το σχέδιο διαχείρισης ε, εδώ στην Επιτροπή Αναφορών. Προτείνω λοιπόν να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορή και να περιμένουμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το αν αρκεί το σχέδιο διαχείρισης ή όχι. Εάν αρκεί μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά. Εάν όχι απαιτούνται και άλλα μέτρα. Να παραμείνει ανοιχτή μέχρι να λάβουμε την απάντηση της Κομισιόν. Αυτή είναι η πρότασή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι τίνετε να συμφωνήσετε με την πρόταση αυτή. Θα ήθελα να προτείνω μια ελαφρά τροποποίηση. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε τη βοήθειά μας. Να στείλουμε λοιπόν επιστολή προς την γαλλική κυβέρνηση, στην οποία να ρωτάμε σχετικά με το σχέδιο δράσης και με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι χθε κατά την συνεδρίαση των συντονιστών λάβαμε απόφαση και θα εξεταστεί το θέμα αυτό. Μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Αφήνουμε ανοιχτή την αναφορά. Στέλνουμε επιστολή προς τις γαλλικές αρχές. Στηρίζουμε έτσι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό όταν θα έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Μπορείτε να συμφωνήσετε με την πρόταση αυτή. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τώρα μια σειρά αναφορών για τους λύκους. Πρόκειται για το τελευταίο ζήτημα που θα συζητήσουμε σήμερα. Θα Συζητήσουμε λοιπόν την αναφορά 1771 κάθετο 2013 του Λουίς Μικέλ Ντομίνγκες Μενσία της Ισπανικής Ιθαγένειας σχετικά με την οδηγία για τους οικοτόπους και την προστασία του λύκου της Ιβηρίας. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι παρόν ο, ε, αναφέρον. Α, όχι, είναι παρόν. Δίνω το λόγο στην αναφέρουσα. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ το Σύλλογο Λόμπο Μάρλι για την προστασία του λύκου της Ιβηρικής Χεροσονήσου. Πριν από ένα χρόνο υπερασπίστηκαμε εδώ την ανάγκη, την επίγουσα να προστατευτεί ο λύκος, ο Ιβηρικός λύκος και καταγγείλαμε τις παρανομίες της Ισπανικής κυβέρνησης. Εν τω μεταξύ έχουν υπάρξει αλλαγές. Η Ισπανική κοινωνία δείχνει όλο και περισσότερο ότι απορρίπτει την άσκοπη και άχρηστη θανάτωση των λύκων, ενώ οι αρνητικές συνέπειες του υφιστάμενου συστήματος ε, γίνονται όλο και πιο εμφανείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν δείχνει ότι την ενδιαφέρουν αυτές οι αλλαγές, γιατί στην ανακοίνωση των μελών ε, δικαιολογεί την πρόθεσή της να κλείσει αυτή την αναφορά. Και αυτή η επιστολή είναι αντίγραφο της επιστολής που μας έστειλε το 2015, που είχε κατάφορα λάθη, τα οποία επαναλαμβάνονται στην νέα εκδοχή της επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και έλλειψη ενδιαφέροντος. Δεν δικαιολογούνται όλα αυτά. Θέλουν να διατηρηθεί ένα σύστημα το οποίο πλήττει την και μάλιστα αυξάνει τα προβλήματα των κτηνοτρόφων. Ορίστε λοιπόν, θα σα μιλήσω για κάποια από τα πιο σοβαρά λάθη τη ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επίστολη επιβεβαιώνει ότι ο ευηρικό λύκο ζει σε θετικέ ευνοϊκέ συνθήκε διατηρείται ε, στην ορεινή περιοχή. Αν δούμε όμω ε, την έκθεση τη Ισπανική κυβέρνηση, βλέπουμε ότι ο πληθυσμό των λύκων δεν υπάρχει ε, στην έκθεση που συνοδεύει το χάρτη. Και μάλιστα αυτός, αυτό το λάθος ήδη βρισκόταν ε, και υπήρχε στο χάρτη του 2015, άρα δεν το ξαναείδαν από τότε. Δεύτερον, σύμφωνα με αυτό το χάρτη, ο πληθυσμός των λύκων στην Ανδαλουσία είναι 42-49 ζώα και επαναλαμβάνει τα δεδομένα του 2015. Όμως έχουμε πιο πρόσφατες πληροφορίες και στοιχεία του 2017 από τον βιολόγο Χουάν Κάρλος Μπλάνκο, τα οποία δείχνουν αυτά τα στοιχεία ότι ο λύκος στην Ανδαλουσία έχει εξαφανιστεί κατά πάσα πιθανότητα. Το να αποφάσεις λοιπόν με τόσο απειρχαιωμένες πληροφορίες και όχι επικυροποιημένες είναι απαραίτητο απαράδεκτο. Και υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στην προστασία του λύκου από τη μία περιοχή στην άλλη ε, και ε, ε, οι διαφορές αυτές είναι που κάνουν το λύκο στην Ανδαλουσία να είναι πάρα πολύ απομονωμένος, να έχει σχεδόν εξαφανιστεί και αν υπάρχουν κάποια ζώα, κάποιοι λύκοι που ζουν ακόμα εκεί και δεν έχουν εξαφανιστεί, είναι τόσο μικρό το γενετικό του υλικό που ε, ο πληθυσμός τους θα αδυνατήσει, το γονιδίωμά τους θα αδυνατήσει και τελικά θα εξαφανιστούν. Έχουμε το έργο LIFE για τον λύκο της Ανδαλουσίας και αυτό το σχέδιο έχει, έχει πεταχτεί στα σκουπίδια τελικά η έλλειψη γενετικής ποικιλομορφίας πλήττει ε, τον πληθυσμό του λύκου σε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο και το πρόβλημα αυτό θεωρεί ότι και σύμφωνα με το πρόβλημα αυτό θα αργήσουν πολύ, θα αργήσει πολύ να αυξηθεί ο πληθυσμός ε, των λύκων. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία, έχουμε κατεξαίρεση θανατώσεις λύκων στην νότια, στη νότια όχθη, από κάτω από τον ποταμό Ντουέρο, όπου εκεί προστατεύεται αυστηρά ο, ο λύκος. Υποτίθεται ότι ε, σκοτώνονται μόνο τα προβληματικά ζώα και όταν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική και ότι όταν σκοτώνονται αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την διατήρηση του πληθυσμού. Όμως η αλήθεια είναι διαφορετική, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Έχουμε στείλει βίντεο στην Επιτροπή που δείχνει ε, πώς εγκρίθηκε η θανάτωση δύο λύκων σε περίπτωση κατά την οποία δεν εκπληρούνταν κανένα από τα προαπαιτούμενα και δεν υπήρχε καμία ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο. Επομένως αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν στέκουν επιστημονικά και δεν έχουν την αποδοχή της κοινωνίας. Η σημερινή τάση των βιολόγων αυτή τη στιγμή είναι ενάντια στον έλεγχο των σαρκοφάγων ζώων του πληθυσμού τους διά της επιλεκτικής θανάτωσης. Έχουμε το περιοδικό Journal of Mammalogy, το περιοδικό για τα θηλαστικά και έχουμε εκεί μια εργασία σχετικά. Ε, αυτό, ε, σύμφωνα με τους επιστήμονες, η θανάτωση μεμονωμένων ζωών δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στον πληθυσμό του. Ε, παρακαλώ τους κυρίους τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερωθούν για την επιστημονική επικυρότητα και την επιστημονική πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα... η ιδέα ότι αν σκοτώσουμε δυο-τρεις λύκους η τοπική κοινωνία θα ανεχθεί περισσότερο να υπάρχουν άλλοι λύκοι και να διατηρηθεί ο πληθυσμός τους είναι μια ιδέα εσφαλμένη. Αντιθέτω, ο, ο κόσμος πιστεύει ότι αν έρχεται και η ίδια η κυβέρνηση για να σκοτώσει ε, λύκους, τότε αυτό σημαίνει ότι το ζώο δεν έχει καμία αξία και άρα μπορεί να το κάνει και η ίδια και μπορεί να το κάνει ο καθένας. Τα έχουμε ζήσει αυτά και στην Αστούρια σε άλλη ε, περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, σύσσωμη η ισπανική κοινωνία εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από την νομοθεσία είτε την εθνική είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει φανεί με τις τεράστιες διαδηλώσεις υπέρ της διατήρησης του πληθυσμού του λύκου στη Μαδρίτη το 2016-2017. Όλο και περισσότερο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα φαίνονται ως ε, μινάρια του παρελθόντος και όχι εργαλείο προόδου. Ο κύριος Μάρκο Τσιπριάνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ έχουμε δύο αναφορές. Την πρώτη τη συζητήσαμε τον Νοέμβριο του 2015 και κάναμε κάποια σχόλια τα οποία ισχύουν ακόμη. Η δεύτερη αναφορά είναι καινούρια. Για το ίδιο θέμα όμως. θέτει και κάποια νέα στοιχεία, το θέμα της διαχείρισης. Η διαχείριση, ακόμη και όταν επιτρέπεται βάσει της οδηγίας, δεν θα πρέπει να είναι συνώνυμη με τη διαχείριση του κυνηγιού. Η διαχείριση δεν είναι ταυτόσιμη με το κυνήγι. Αυτό λέει η αναφορά και εμείς είμαστε σύμφωνοι. Η διαχείριση είναι ευρύτερος όρος από το κυνήγι. Εξάλλου αυτό δεν είναι μόνο η γνώμη μας, αυτό αποτυπώνεται και στα σχέδια διαχείρισης και στην Ισπανία και σε άλλα κράτη-μέλη. Η διαχείριση μεγάλων σαρκοβόρων μπορεί να περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Παραδείγματο χάρη θέματα διαχείρισης οικοτόπων, εξασφάλιση επαρκούς δασοκάλυψης για τους λύκους, προστασία ευαίσθητων περιοχών του οικοσυστήματος, σημεία στα οποία ε, φέρνουν τα μικρά τους ε, οι λύκοι. Προσπαθούμε να μειώσουμε τη θνησιμότητα, να μειώσουμε τον κατακαιρματισμό, να μην ε, κατακαιρματίζονται αυτοί οι κότοποι από υποδομές μεταφορών εξασφαλίζεται και επαρκής λία για τους λύκους, ε, ελάφια, αγριογούρουνα κλπ. Διαχείριση σημαίνει και διαχείριση συγκρούσεων, δηλαδή αντιμετώπιση όλων των θεμάτων τα οποία προκύπτουν λόγω της παρουσίας των λύκων. Αυτό σημαίνει υποστήριξη και βοήθεια προς όσους φύγονται με διάφορα μέτρα. Ε, διαχείριση συμπεριλαμβάνει και την έρευνα και συγκέντρωση δεδομένων για τη διαμόρφωση ορθής πολιτικής. Στοιχεία για τον πληθυσμό, για την περιοχή, για την διατροφή, για την επίπτωση των ζώων την επίπτωση επί των ε, ζώων κτηνοτροφίας, διάδοση του είδους, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αν το είδος όμως αυτό αναφέρεται στο παράρτημα 5 της ε, οδηγίας για τους οικοτόπους, διαχείριση επιτρέπεται να περιλαμβάνει και τη θύρα. Στο βαθμό βέβαια που μιλάμε για βιώσιμη θύρα. Συμβατεί με την διατήρηση των ειδών. Και συγκεκριμένα για την κατάσταση στην Ισπανία, για το λύκο βορείου του ποταμού Ντουέρο, όπου ζει το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του μεγάλου πληθυσμού λύκων, σύμφωνα με την οδηγία για τα οικοσυστήματα, ο πληθυσμός των λύκων μπορεί να είναι αντικείμενο θύρας και σε άλλες περιοχές άλλων κρατών μελών, στην Ελλάδα σε κάποια σημεία, στη Φινλανδία, στη Σλοβακία, σε, στις χώρες της Βαλτικής, στην Πολωνία, επιτρέπεται η θύρα ορισμένων ειδών λύκων. Η οδηγία λέει ότι επιτρέπεται η θύρα, δεν λέει ότι πρέπει να ισχύει η θύρα, επειδή η οδηγία λέει ότι υπάρχει δυνατότητα, ορισμένες χώρες ε, ε, επιλέγουν να το αντιμετωπίζουν ως πλήρως προστατευόμενο είδος. Απλώς επιτρέπεται η θύρα, δεν επιβάλλεται. Βορείως του ποταμού του Αέρο επιτρέπεται λοιπόν ε, το κυνήγι εφόσον υπάρχει επαρκή διατήρηση αυτού του είδους λύκου. Σύμφωνα με τις εκθέσεις που έχει υποβάλει η Ισπανία στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 17 της Οδηγίας για τα οικοσυστήματα, ο λύκος φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια ευνοϊκή κατάσταση. Μιλάμε για μεγάλο πληθυσμό, 2.500 άτομα. Στο Νότο, στη Σιέρα Μορένα, υπάρχει μια εξαίρεση και το αναγνωρίζουν αυτό οι Ισπανικές αρχές. Και αυτό αποτυπώνεται στην έκθεση βάσει του άρθρου 17. Η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση και τις εξελίξεις στην Σιέρα Μορένα και είναι συνεχώς σε επαφή με τις Ισπανικές Αρχές. Εν κατακλείδη. Οι αναφέροντες ζητούν να αλλάξουν τα παραρτήματα της οδηγίας και να επεκταθεί το αυστηρό καθεστώς προστασίας σε ολόκληρη την Ισπανία, δηλαδή και βορείως του ποταμού Ντουέρο. Μάλιστα, Έχουμε λάβει και αιτήματα από την Ισπανία να αλλάξουν τα παραρτήματα κατά τον αντίθετο τρόπο. Από την Ισπανία μας έχουν στείλει αιτήματα να μην υπάρχει καθόλου αυστηρό καθεστώς βορείως του ποταμού αέρο. Η θέση της Επιτροπής είναι ότι το τρέχον νομικό πλαίσιο το θεωρούμε κατάλληλο και ορθό και δεν θα προτείνουμε αλλαγές για τις οδηγίες και για τα παραρτήματα. στα πρόσφατα συμπεράσματα του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας, το πόρισμα ήταν ακριβώς αυτό. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι σωστό το νομικό πλαίσιο, παρέχει επαρκή ευελιξία στις εθνικές αρχές και συνάδει προς το στόχο του να διατηρήσουμε ευνοϊκό καθεστώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πρωτού να ανοίξουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι χθες, κατά την συνάντηση των συντονιστών, συζητήθηκε το θέμα αυτό, διότι λάβαμε σχετικές πληροφορίες. Έχουν αναθέσει λοιπόν την μελέτη της κατάστασης που θα διαρκέσει κάποιους μήνες. Δεν μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε ακόμα την αναφορά. Περιμένουμε στοιχεία από την Ισπανική κυβέρνηση, καθώς και τα αποτελέσματα της δικής μας αξιολόγησης. Θα συζητήσουμε λοιπόν το θέμα, δεν θα μπορέσουμε όμως να το κλείσουμε. Κύριο κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους αναφέροντες από την Ισπανία για την υποβολή αυτής της αναφοράς. Και δεν είναι και μόνο τους. Πρόσφατα Πάρα πολλοί πολίτες στην Ισπανία διαδήλωσαν στη, στη Μαδρίτη ζητώντας την προστασία του ιβυρικού Λύκου. Ο Λύκος είναι ένα είδος ε, ε, ζωικό, ε, ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση πολλών και διαφορετικών οικοσυστημάτων στην Ισπανία. Είναι απόλύτω εφικτή η συνύπαρξη του Λύκου με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, με επεκτεταμένη και αηφόρο και βιώσιμη κτηνοτροφία. Είναι επίσης ο λύκο πόλος έλξης για τη φυσικότητα ενό τοπίου, κάτι το οποίο το κάνει εξαιρετικά ελκυστικό τουριστικά δεν βλάπτει η παρουσία του υλικού καμία ανθρώπινα ε, δραστηριότητα. Όμως πρέπει ε, σύμφωνα με την νομοθεσία και τις αντίστοιχες οδηγίες να μπορεί το είδος το επαπειλούμενο να ζει σε ευνοϊκές και θετικές για την εξέλιξή του συνθήκες. Ε, αυτή τη στιγμή στην Ισπανία δεν εκπληρούνται τα προαπαιτούμενα ε, στα άρθρα 14 και 16 της σχετικής οδηγίας. Στην αυτόνομη κοινότητα της Καστήλης Λεών, στην περιοχή Άβυλα, οι αρχές κήρυξαν την περιοχή ελεύθερη λύκων. Αυτό δεν είναι βιώσιμη διαχείριση της διαφοράς. Δεν μιλούμε για διατήρηση, μιλούμε για εξάλληψη, για εξόντωση από πλευρά Ισπανικών αρχών και θέλω να υπενθυμίσω ότι αυτέ οι δράσει στην Ισπανία αντίκυνται στην ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και εμεί, ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ω Επιτροπή Αναφορών, ω μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Πρέπει να αναλάβουμε δράση για, το, για τη τήρηση της και για την επαρκή ε, προστασία και διατήρηση του πληθυσμού των λύκων. Χαίρομαι που θα παραμείνει ανοιχτή αναφορά και ελπίζω ότι θα έχουμε μια έκθεση που θα αναδεικνύει τις κακές πρακτικές στην Ισπανία και ε, θα προβάλλει εναλλακτικέ λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, επόμενος ομιλητή Αράντσο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη γιατί καθυστέρησα, αλλά έρχομαι από την Επιτροπή Ενέργειας και Βιομηχανίας. Θέλω να ευχαριστήσω την οργάνωση Λόμπο Μάρλι γιατί θέτει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το θέμα που το τόσο ενδιαφέρον. Ε, πρέπει να, να πράξουμε όλοι τα δέοντα για να βοηθήσουμε στην επιβίωση αυτού του είδους και στην προστασία του. Ο, ο λύκος έχει υψηλή κυνηγητική αξία, ε, ε, ε, είναι μέρος του συλλογικού μου ασυποσυνείδητου και η διατήρησή του είναι απολύτως απαραίτητη. Ε, ελέγχει λόγω της δράσης του το πληθυσμό άλλων ειδών, τα οποία αν δεν υπάρχει ο λύκος, τα οποία τα τρώει στη διατροφική αλυσίδα, θα μας κατακλείσουν. Επομένως βοηθάει πάρα πολύ τον κύκλο ζωής. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι το κυνήγι του λύκου και η θανάτωση μεμονωμένων ζώων υποτίθεται για τη ε, ε, διατήρηση του είδους ε, οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα. Σκοτώνονται κάποιοι λύκοι, αλλοιώνεται το κοινωνικό σύστημα της αγέλης των λύκων που λειτουργεί με συγκεκριμένη πυραμίδα και πλήττονται οι κυνηγητικές ιδιότητες του ζώου και άρα υπάρχει πλήρη διατάραξη του κύκλου ζωής και της διατροφικής αλυσίδας στη φύση. Και μετά πρέπει να αντιμετωπίσουμε άλλα προβλήματα. Βεβαίω πρέπει να αποζημιώσουμε ή να λύσουμε το πρόβλημα των κτηνοτρόφων που χάνουν ζώα. Όμω δεν, θα το λύσουμε σκοτώνοντα λύκου. Σκοτώνοντα λύκου πλήττουμε άλλου οικοτόπου και άλλα βιοσυστήματα. Ε, μπορούμε να στηρίξουμε αυτού του ανθρώπου, του κτηνοτρόφου, για τα προβλήματα, ε, να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρο, από ό,τι φαίνεται, χθε. Ε, οι συντονιστές ζήτησαν την εκπόνηση και σύνταξη περιεκτικής ολοκληρωμένης μελέτης. Υπάρχει ένας νέος γύρος επικοινωνίας μεταξύ Ισπανικών Αρχών, Ισπανικής Κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με βάση όλα αυτά, κρατούμε την αναφορά ανοιχτή προτείνω και μόλις έρθουν νέα στοιχεία θα επανέλθουμε. Εάν συμφωνείτε, πάμε... Προχωρούμε 2348 του 2014. Άντολφ Γουίτ από την Γερμανία. 2348 αναφορά του 2014 για το πληθυσμό των λύκων στη Γερμανία. Ο αναφέρον δεν είναι παρόν, εξ όσων γνωρίζω, στην κάτω Σαξονία. Ο κύριος Μάρκο Τσιπριάνη έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ αναφέρον μας ζητά κατά βάση να αλλάξουμε το παράρτημα της οδηγίας για τα οικοσυστήματα και να μην υπάρχει αυστηρή προστασία του λύκου στη Γερμανία και να επιτρέπεται η θύρα. Και αυτή η αναφορά είχε συζητηθεί εδώ το Δεκέμβριο του 2015. Και συνεχίζουν να ισχύουν τα σχόλια που είχαμε κάνει τότε. Το μόνο σημαντικό νέο στοιχείο είναι το συμπέρασμα της αξιολόγησης ε, της οδηγίας ε, για το περιβάλλον βάσει του εγγράφου της Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου του 2016. Το πόρισμα λοιπόν από την αξιολόγηση καταλληλότητας είναι ότι οι οδηγίες για τα οικοσυστήματα των πτηνών παραμένουν ενισχύ και παρέχουν επαρκή ευελιξία στα κράτη-μέλη ώστε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα υλοποίησης. Η Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει κατά την υλοποίηση και θα βοηθήσει διότι και τώρα διαμορφώνουμε ένα σχέδιο δράσης για την βελτίωση της υλοποίησης. Επομένως, η, οδηγία, η Επιτροπή συγγνώμη, δεν προτίθεται να προτείνει αλλαγές ούτε για την οδηγία ούτε για τα παρατήματα αυτής. Αυτό σημαίνει ότι ο λύκος στη Γερμανία θα παραμείνει στο παράρτημα 4, δηλαδή αυστηρά προστατευόμενα είδη. Όμως, αυτό το θέμα του παραδείγματος 4 και του παραδείγματος 5 δεν είναι το πραγματικό ζήτημα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Η συνύπαρξη είναι το πρόβλημα. Συνύπαρξη σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά τα είδη, με αυτά τα μεγάλα σαρκοβόρα. Θα πρέπει να μάθουμε να μοιραζόμαστε τη φύση με αυτά τα ζώα και με άγρια ζώα, δηλαδή περιλαμβανομένου του λύκου. Και αυτά υπάρχουν και στο παράρτημα 4 και στο παράρτημα 5. Το ευνοϊκό καθεστώς ε, συντήρησης που είναι στόχος της οδηγίας πρέπει να επιτευχθεί και με το παράρτημα 4 και με το παράρτημα 5. Η συνύπαρξη είναι μια πρόκληση που σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε σε μέτρα πρόληψης για να αποφύγουμε απώλεια ζωής, να πρέπει να βελτιώσουμε την πληροφόρηση, να βελτιώσουμε το διάλογο με τις κατηγορίες που πλήττονται και με, το, με την κοινή γνώμη γενικότερα. Και το κάνουν αυτό στην Σαξονία, γιατί περί της Σαξονίας πρόκειται στην αναφορά αυτή. Σύμφωνα με την επιστολή αυτή που εστάλει στην Επιτροπή Αναφορών από τις τοπικές αρχές της Αξονίας πέρυσι τον Ιούλιο, εξηγούν ότι υποστηρίζουν τους κτηνοτρόφους για την πρόληψη και με αποζημίωση ζημιών, υποστηρίζουν την έρευνα, την παρακολούθηση, εκστρατείες ενημέρωσης και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας στέλνουν, η προσέγγισή τους θεωρείται επιτυχημένη έχει καταφέρει να κρατά σε χαμηλά επίπεδα τις ζημίες, τις απώλειες, παρότι αυξάνεται ο πληθυσμός των λύκων στην περιοχή και είναι επιτυχημένη αυτή η εκστρατεία διότι η ε, πλειοψηφία των κατοίκων στη Σαξονία είναι υπέρ των μέτρων αυτών σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν γίνει. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την ορθή προσέγγιση της Σαξονίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται να είναι καλύτερη η κατάσταση λοιπόν σε αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα. Γιάχ. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει και στον αναφέροντα να το αναφέρουμε ότι ε, κατά την Επιτροπή ε, πρέπει να υπάρχει ευελιξία πρέπει να υπάρχει ευελιξία σε κάθε κράτο μέλο και είναι ικανοποιημένη η Επιτροπή από την ευελιξία που υπάρχει και από ό,τι φαίνεται από αυτό που μα λέει και η Επιτροπή είναι θετικά ε, τα μέτρα. Έχουμε ακολουθήσει εκστρατείε ενημέρωση τα τελευταία δέκα χρόνια. Έχει αυξηθεί ο πληθυσμό των λύκων. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Τι κάνουμε με λύκους που έχουν παραπτωματική συμπεριφορά, γιατί δεν μπορούμε να τους σκοτώσουμε όλους. Ε, τι κάνουμε όταν ένας λύκος ε, δεν ακολουθεί την σωστή συμπεριφορά. Ε, υπάρχουν θέματα τα οποία δεν μπορεί να μας τα απαντήσει η Επιτροπή. Είναι θέματα που θα πρέπει η περιφέρεια να τα απαντήσει. Να κλείσουμε την αναφορά λοιπόν, αλλά να απαντήσουμε στον αναφέροντα και να πούμε ότι στην κάθε περιφέρεια, στη συγκεκριμένη περιφέρεια της Γερμανίας, θα πρέπει ε, να ε, υπάρχει φιλική συνύπαρξη του ανθρώπου με το λύκο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε σωστά συστήματα διαχείρισης. Και έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι θέματα επικουρικότητας αυτά γιατί στις Βρυξέλλες πού να ξέρουν πόσους λύκους έχει η Σαξονία. Πρέπει η Σαξονία να το κρίνει και να το αποφασίσει και να το τηρήσει. Προτείνω λοιπόν να κλείσουμε την αναφορά ε, εξηγώντα ε, στον αναφέροντα ότι πρέπει να στραφεί ενδεχομένω στις τοπικές αρχές για να συζητήσει το θέμα αυτό περαιτέρω, διότι υπάρχει ευελιξία για τα κράτη-μέλη και ότι είμαστε ικανοποιημένοι, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει επομένως ε, άμεση ανάγκη να ληφθούν κάποια μέτρα από αυτού και να αλλάξει κάτι. Τουλάχιστον για αυτό που συζητάμε για τη Σαξονία. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι από ό,τι μας είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ικανοποιημένη με τα ευρήματά τους. Ο Πίτερ Γιά προτείνει να το κλείσουμε το θέμα και να στείλουμε αντίστοιχη επιστολή που θα το εξηγούμε. Ο κύριος Εκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που μπορούμε να κλείσουμε μια αναφορά και χαίρομαι που και η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τήρει μια σωστή στάση όσον αφορά την συνύπαρξη με το ΛΥΚΟ. Νομίζω ότι υπάρχει μια παράλογη σχέση όσον αφορά την συνύπαρξη ανθρώπου και λίγου χθε. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος συζητούσαμε τα θέματα αυτά και είπε ένας συνάδελφος ότι οι μαμάδες φοβούνται να αφήσουν τα παιδιά τους να βγουν να περπατήσουν. Παραλογισμοί δηλαδή. Θα πρέπει να έχουμε κατά ότι μέχρι τώρα στη Γερμανία Ούτε ένας άνθρωπος δεν ε, έχει πέσει ε, θύμα επίθεσης ε, λύκου. Ξέρετε όμως πόσα θύματα έχουμε από επιθέσεις κυνηγών. Σαράντα. Έχουμε θύματα από κυνηγού που περιπλανώνται αμέριμνοι στη φύση. Ίσως λοιπόν θα ήταν σκόπιμο να κάνουμε μια σχετική μελέτη. Ευχαριστώ πολύ. Άρα η πρόταση του Πέτα Γιάχ και την πρόταση την οποία θα αποδεχθούμε είναι να κλείσουμε την αναφορά αυτή. Η επόμενη αναφορά είναι η παριθμόν 11 του 2015 της Ιωάννα Παρίκα Αλτενστέτ, Σουηδικής Ιθαγένειας, σχετικά με το κυνήγι λύκων στη Σουηδία. Δεν είναι παρούσα η αναφέρουσα. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λίντα Νίρεν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα του κυνηγιού του λύκου στην ε, Σουηδία είναι ένα θέμα πολύπλοκο. Καταρχάς, ε, πρέπει να γνωρίζουν ε, οι άνθρωποι ότι οι αποφάσεις που τους επηρεάζουν λαμβάνονται από ανθρώπους που γνωρίζουν την κατάσταση. Η αρχή της επικουρικότητας θεσπίζεται και στη συνθήκη. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι εθνικοί δικαστές είναι καταρχάς αρμόδιοι για την διασφάλιση της σωστής εφαρμογής ε, της ε, νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα κράτη-μέλη. Εάν όμως υπάρχουν εμπόδια στην πρόσβαση προς τους δικαστές, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει για να διασφαλίσει την σωστή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Και αυτό συνέβη στη Σουηδία, διότι το 2010 όταν ξεκίνησε το κυνήγι με άδειε, οι περιβαλλοντικέ μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, ούτε, ήταν, ε, ούτε συμμετείχαν στη διαδικασία, ούτε είχαν τη δυνατότητα να ασκήσουν έφεση. Έτσι λοιπόν ε, υπέβαλαν ένσταση στην Κομισιόν διότι δεν είχαν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και δεν είχαν και άλλη λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία επιπαραβάση μέχρι το 2013 που ε, ε, επέτρεπε πια το σουηδικό σύστημα πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και έτσι επέτρεπε την ε, άσκηση έφεσης για τις αποφάσεις σχετικά με το κυνήγι λύκου στα εθνικά δικαστήρια. Ωστόσο, το 2014 η Σουηδία αποφάσισε από την κεντρική διοίκηση στην ε, Στοκχόλμη να ε, μεταφερθεί η αρμοδιότητα στις νομαρχίες όπου πραγματοποιείται το κυνηγή Αυτό από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι προβληματικό διότι έτσι λαμβάνονται οι αποφάσεις πιο κοντά στους πολίτες. Έτσι όμως η Σουηδία ε, είχε, επέβαλε περιορισμό στην πρόσβαση των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη δικαιοσύνη λόγω των ε, κανόνων που ίσχυαν σχετικά με τι αποφάσεις και αυτή η απόφαση δεν ε, συνάδει με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και γι' αυτό ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία επιπαραβάσης σχετικά με την πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν είχαμε δύο διαδικασίες επιπαραβάση, μία που αφορούσε την πρόσβαση στη διαδικασία και την άλλη που αφορούσε το κυνήγι λύκου αυτό καθ' αυτό. Ε, η διαδικασία επί παραβάση για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη ήταν σημαντική, οδήγησε σε τροποποίηση της Σουηδικής ε, νομοθεσίας, το οποίο σημαίνει ότι από τον Απρίλιο του 2016 οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν πάλι το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση ε, στα διοικητικά δικαστήρια της Σουηδίας και έτσι μπόρεσε να κλείσει αυτή η διαδικασία επί παραβάση. Τώρα έχουμε πια τις ε, εφέσεις ε, των περιβαλλοντικών με κυβερνητικών οργανώσεων που επέτρεψαν ε, στην, στο Διοικητικό Δικαστήριο της Σουηδίας να λάβει απόφαση σχετικά με το κυνήγι λύκου που εγκρεμεί από το 2010 και πρόκειται για το πιο υψηλοπάθμιο δικαστήριο στην Σουηδία για το θέμα αυτό. Όσον αφορά λοιπόν τα... το κυνήγι, ε, η απόφαση αυτού του υψηλού δικαστηρίου δεν να πάντα με ε, αποφάσεις πιο χαμηλό βαθμών δικαστηρίων και γι' αυτό ε, θα πρέπει να εξετάσουμε αναλυτικά την υπόθεση προτού λάβουμε απόφαση για οποιαδήποτε διαδικασία επιπαραβάση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, περνώ το λόγο να μιλήσω για το θέμα αυτό. Φυσικά η υπόθεση αυτή σωστά την χειρίζεται η Κομισιόν Απλά μου δίνετε αφορμή, επειδή συζητούμε το θέμα της προστασίας των λύκων, να θέσω ένα ζήτημα το οποίο αφορά και τους ε, κτηνοτρόφους. Έχω μπροστά μου μία επιστολή των κτηνοτρόφων της περιοχής Ορεινής Τριχονίδας. Είναι στην περιοχή της Ετωλοκαρνανίας με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 2016 στην Ελλάδα. Οι κτηνοτρόφοι λοιπόν αυτοί έχουν αποστείλει υπόμνημα στο Υπουργείο Γεωργίας, διαμαρτυρώμενοι ότι στην περιοχή τους τα κοπάδια τους δέχονται συνεχείς επιθέσεις από λύκους και έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Μάλιστα καταγγέλουν ότι οι οικολογικές οργανώσεις αφήνουν στην περιοχή τους ελεύθερους λύκους στο πλαίσιο της οικολογικής προστασίας όπως λένε. Άρα λοιπόν εκτός από τις πλευρές που αναφέρθηκαν σωστά από τους συναδέλφους για το ρόλο που παίζουν οι λύκοι στην οικολογική ισορροπία και το οποίο σωστά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με μια νομοθεσία προστασίας του, των ζώων αλλά ταυτόχρονα και με ένα ελεγχόμενο κυνήγι. Ε, ήθελα να θέσω υπόψη της Επιτροπής σας ότι σύντομα θα αντιμετωπίσουμε αιτήματα από την άλλη πλευρά. Δηλαδή υπάρχουν ε, μια σειρά κτηνοτροφικές οργανώσεις. Αυτό εδώ το υπόμνημα το υπογράφουν 900 κτηνοτρόφοι και οι οποίοι αυτό που ζητούν είναι να πάρουν κάποιες αποζημιώσεις. Διότι η ισορροπία σε όλα τα θέματα, όπως είναι και η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία των ζώων, η προστασία των άγριων ζώων, η προστασία του λύκου, οπωσδήποτε πρέπει να σταθμιστεί και με κάποιες αποζημιώσεις απέναντι στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι υφίστανται τεράστιες ζημιές στα κοπάδια τους. Αυτή δε η επιστολή την οποία σας αναφέρω των κτηνοτρόφων της ορεινής ναυπακτίας ε, και της ετολοκαρνανιές είναι ενδεικτική του τι συμβαίνει. Απ' τη μια πρέπει να υπάρξει προστασία, απ' την άλλη να υπάρξει και απαγόρευση στις οικολογικές οργανώσεις να αφήνουν ελεύθερους λύκους σε μια σειρά περιοχές και επίσης να ληφθεί υπόψη και ο τρόπος με τον οποίο θα προστατευτούν και οι ίδιοι κτηνοτρόφοι. Το λέω αυτό λοιπόν για να το έχει υπόψη η Κομισιόν, μια και ορθώς ακούει τα ζητήματα αυτά, αλλά να σταθμίσει και τα συμφέροντα γιατί σύντομα βλέπω να έχουμε αναφορές εδώ από την άλλη πλευρά. Ότι δηλαδή πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα προστασίας αυτών των ίδιων των κτηνοτρόφων που ζουν σε αυτές τις ορεινές περιοχές, ιδίως στην Ελλάδα που έχει φτωχοποιηθεί αυτή τη στιγμή ο κτηνοτρόφος και λόγω της πολιτικής των μνημονίων και άρα είναι ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει να το λάβει υπόψη η Επιτροπή μας, δηλαδή να έχουμε ορθά την εφαρμογή της οικολογικής νομοθεσίας, αλλά να δούμε και την άλλη πλευρά Επομένως συμφωνώ με τις τοποθετήσεις που είχαν προηγουμένως από τον κύριο Γιάρ και άλλους συναδέλφους ότι είναι ένα θέμα επικουρικότητας. Δηλαδή τα ίδια τα κράτη ξέρουν τι συμβαίνει σε κάθε περιοχή. Έχουμε σοβαρά μια νομοθεσία γενική η οποία ορθώς βάζει τους άξονες αλλά πρέπει σε κάθε κράτος να επικρατήσει η αντίστοιχη ευελιξία και το αντίστοιχο Υπουργείο με βάση τα φαινόμενα σε κάθε περιοχή ακόμη και σε κάθε περιοχή, κάθε κράτους, να μπορεί να λάβει μέτρα, ούτω ώστε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην προστασία των άγριων ειδών, όπως είναι ο λύκος, αλλά και στην προστασία της οικονομικής δραστηριότητας, κυρίως των κτηνοτρόφων, και της προστασίας της ζωής. Φυσικά δεν έχουμε επιθέσεις μέσα σε κατοικημένες περιοχές, αλλά έχουμε επιθέσεις σε ορεινές περιοχές, κυρίως σε κοπάδια. Άρα αυτή είναι η δικιά μου παρέμβαση στο θέμα αυτό, ως ένας προβληματισμός για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο Πέτερ. Ναι, να... Το ξανατονίσω, οι δικές μου εμπειρίες ε, και αυτές παίρνουμε εδώ στις Βρυξέλλες, είναι ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται ε, εντατικός διάλογος επιτόπου και το έχω πει και αλλού χωρίς να γίνει κάποια αναφορά, χωρίς να γίνει κάποια αίτηση, δεν γίνεται τίποτα στις Βρυξέλλες. Δεν μπορεί να περιμένει κανείς οι Βρυξέλλες την κατάσταση στην Ελλάδα να μπορεί να την ε, αξιολογήσουμε. Εξαρτόμαστε από την αρχή της επικουρικότητας. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να έχουμε τη στρατηγική, πρώτα να πηγαίνουμε επί τόπου, να βλέπουμε πώς έχει η κατάσταση Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, συνεχίζει να επιτρέπεται η πληρωμή αποζημίωσης στους ε, γεωργούς, ε, να εφαρμόζονται ε, μέτρα προστασίας, αλλά αν δεν λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να συζητώνται. Θα πρέπει να συζητάμε μήπως πράγματι ο αριθμός των λύκων έχει αυξηθεί υπερβολικά. Ε, αλλά οι Βρυξέλλες συχνά κατηγορούνται ότι αποφασίζουν ε, τα πάντα. Αλλά όταν αποφασίζουν οι περιφέρειες, τότε τα παράπονα φτάνουν στις Βρυξέλλες. Εμάς ε, ξαναεμφανίστηκαν οι λύκοι μετά, πριν από 100 χρόνια και έχουν διχάσει τους πολίτες. Γι' αυτό άλλωστε λάβαμε και την ε, σχετική αναφορά. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω τις περιφέρειες να φροντίσουν για καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες και να χρησιμοποιήσουν το περιθώριο που τους επιτρέπει ο Ευρωπαίος Νομοθέτης. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ευρύτερο περιθώριο από ό,τι νομίζουν και οι δύο πλευρές. Και αν οι Βρυξέλλες πούνε αυτό δεν το δεχόμαστε καθόλου, τότε να συνομιλήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει πάντα και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Εύη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πάρω το λόγο για το θέμα αυτό, ε, κάνοντας ένα γενικότερο σχόλιο. Αυτή η αναφορά η Σουηδική έχει να κάνει με τα μέτρα διατήρησης και προστασίας ε, και έχει να κάνει και ε, με τη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να, ε, για να υπάρξει μια ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ ανθρώπου και λύκου κατά πάσα πιθανότητα είναι απαραίτητο να ε, δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές και να εμπνευστούμε από αυτές. Προσωπικώς καταγγέλλω το κυνήγι. Θεωρώ ότι το 2017 πρέπει να εξαφανιστεί αυτή η πρακτική. Δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος του σχεδίου διαχείρισης των ε, εδαφών. Εγώ νομίζω ότι είναι μια δραστηριότητα εξωφρενική σήμερα. Μπορεί να υπάρξουν και άλλες λύσεις. Και θέλω νομικά να αναφερθώ στο θέμα των αγριογούρουνων των αυτόχθονων ειδών που έρχονται από άλλα μέρη της Ευρώπης. Είναι πρόβλημα, γιατί έχει αυξηθεί ο πληθυσμός τους. Πολύ συχνά ο άνθρωπος παίρνει αποφάσεις που τελικά είναι κακές και αυτές ε, πλήττουν το περιβάλλον στο οποίο διαβεί. Και δημιουργούνται και τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκε και ο ε, συνάδελφος κ. Μαριάς. Σαφέστατα υπάρχει οικονομικός αντίκτυπος ε, στη γεωργική παραγωγή, την τοπική, στην κτηνοτροφική παραγωγή. Και πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Νομίζω ότι το κυνήγι ως επίσημο μέτρο δεν θα πρέπει να υφίσταται, να, δηλαδή να, ε, να επιτρέπουμε το κυνήγι ως μέτρο ελέγχου του πληθυσμού. Στην Ιταλία επανενεργοποιήθηκε η αδειοδότηση του κυνηγιού με αδειοδότηση συγκεκριμένων μεμονωμένων ζώων που ε, μπορεί ένας κυνηγός να σκοτώσει. Αυτό θέλησε η Ιταλική κυβέρνηση να κάνει, αλλά ευτυχώς καταφέραμε να σταματήσουμε να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την τρέλα. Τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της επικράτειας, της περιοχής, της εκάστοτε, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη του στην ειρηνική συμβίωση ανθρώπου και λύκου, χωρίς να προσφεύγουμε σε αυτή τη βάρβαρη δραστηριότητα, η οποία δεν έχει κανένα νόημα πλέον σήμερα, από τη στιγμή που υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις και αυτές οι πρακτικές μπορούν να ενισχυθούν και να διαδοθούν περαιτέρω. Να εθετήσουμε τις καλές πρακτικές γιατί υπάρχουν. να τις υιοθετήσουμε εκεί όπου ε, χρειάζεται για να μπει ένα τέλος σε μια δράση η οποία δεν ανήκει πλέον στη σημερινή εποχή. Ευχαριστώ. Ο κύριος καθηγητής Μπρούμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, οι λύκοι ζουν σε αγέλες, είναι κοινωνικά ε, όντα και αν υπάρχει διατάραξη της ομάδας επειδή θα θανατωθεί ένα ή δύο ζώα που ανήκουν στην αγέλη, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες να δημιουργηθεί πρόβλημα στα υπόλοιπα ζώα. Και μάλιστα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να επιτεθούν σε κοπάδια οι υπόλοιποι λύκοι γιατί έχει διαταραχθεί ο κύκλος και η ισορροπία η κοινωνική εντός της αγέλης επειδή έχουν ε, σκοτωθεί κάποια μέλη της. Στις, σε ορισμένες περιοχές στην Ευρώπη Είναι πολύ δύσκολο οι κτηνοτρόφοι να ξέρουν αν τα ζώα τους ε, σκοτώθηκαν από λύκους, κατασπαράχθηκαν ή από ένα είδος σκυλιού το οποίο είναι εξαιρετικά άγριο αλλά δεν ανήκει ε, στο πληθυσμό των λύκων. Βεβαίως εγώ τα ξεχωρίζω αλλά θεωρώ ότι πρέπει νομικά να γίνει διαφορά. Δηλαδή η πολιτεία είναι υπεύθυνη για αυτά τα άγρια σκυλιά και το είδος τους, άρα οφείλει να αναλάβει δράση, ενώ ο λύκος είναι ένα άγριο ζώο που ζει ελεύθερο στη φύση και αυτό είναι κάτι το τελείως ε, διαφορετικό. Και αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε γιατί θα διαμορφώσουν τη στάση μας. Ο Πρόεδρος, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει το θέμα, είναι σε επικοινωνία με, το, με τις Αρχές ε, νομίζω ότι ε, πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ προσωπικώς στηρίζω τη στάση της και στηρίζω και με τους συναδέλφους. Δηλαδή δεν κλείνουμε την αναφορά αυτή τη στιγμή, περιμένουμε το τέλος της διαδικασίας επί παραβάση, στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι προτάσεις ε, των συναδέλφων του κυρίου Μαριά και του κυρίου και θα εξεταστούν από τους συναδέλφους. Αυτό σας ζητώ να κάνετε οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Προχωρούμε λοιπόν, πάμε στην 764 του 2016. Γαλλική αναφορά. Ο κύριος Τσιπριάνη θα πάρει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν είναι παρόντες οι αναφέροντες. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Γαλλία έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης για το λύκο από το 2003 μέχρι το 2018 που αντικαθιστά το προηγούμενο σχέδιο δράσης που ήταν μέχρι το 2012 για να συμφιλιώσει τις ανθρώπινες δραστηριότητες ε, με την παρουσία και την ε, επέκταση του λύκου. Επομένως, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Γαλλίας αφορά τη συνύπαρξη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω συγκεκριμένων δράσεων. Η πιο σημαντική δράση είναι η υποστήριξη με μέτρα προστασίας ε, της κτηνοτροφίας. Η Γαλλία έχει αρκετά σημαντικό προϋπολογισμό για να στήριξει τέτοια μέτρα με τσοπανόσκυλα, ηλεκτρικούς ε, ε, φράχτες, ε, με βοσκούς φύλακες και μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης χρησιμοποιούν και κοινωνικά, κοινοτικά κονδύλια. Δίνουν και αποζημίωση για απώλεια ζωικού κεφαλαίου που φτάνει στα εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στη Γαλλία. Επίσης υποστηρίζουν την έρευνα και παρακολούθηση, την ενημέρωση. Συμμετέχουν ομάδες ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων για την διαχείριση του λύκου. Και το σχέδιο δράσης επίσης προβλέπει και κάποιες παρεκκλήσεις. Ο λύκος είναι αντικείμενο αυστηρή προστασία στη Γαλλία βάσει του παραρτήματος 4, αλλά η οδηγία έχει τη δυνατότητα παρεκκλήσεων, επιτρέπει δηλαδή κάποια άτομα να εξαιρεθούν εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Για να τα υλοποιήσει όλα αυτά η Γαλλία, έχει δημιουργήσει ένα σύστημα σταδιακής απόκρισης. Δηλαδή πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις πριν περάσουμε στο επόμενο στάδιο και πριν επιτραπεί η θανάτωση ατόμων ε, λύκου. Υπάρχουν μέτρα κατάλληλης προστασίας, υπάρχουν μέτρα εκφοβισμού των λύκων χωρίς να τους θανατώσουν. Στη συνέχεια υπάρχουν ε, πυροβολισμοί άμυνας και πυροβολισμοί άμυνας σε μεγαλύτερο επίπεδο μέχρι να φτάσουμε σε πυροβολισμούς οι οποίοι ε, θανατώνουν το λύκο. Ο στόχος αυτού του σταδιακού συστήματος είναι να περιοριστεί η χρήση των παρεκκλήσεων στο ελάχιστο δυνατόν βάσει της αρχής της αναλογικότητας. Κάποιες διοικητικές αποφάσεις ε, που επιτρέπουν τη θανάτωση των ζώων ήταν πολύ αντιφατικές στη Γαλλία. Υπάρχει όμως ένα ορθό ε, δικαστικό σύστημα και αυτές οι εγκρίσεις πολύ συχνά ε, φτάνουν στα εθνικά δικαστήρια με ενστάσεις και οι δικαστές επαληθεύουν το αν όντως πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις οι προϋποθέσεις και του γαλλικού νόμου και βάσει της οδηγίας ε, για τα οικοσυστήματα. Αν δεν υπάρχει δηλαδή επαρκή συναλλακτική λύση, αν ε, δεν υπάρχει αρνητική επίπτωση στο καθεστώς ευνοϊκής προστασίας, μερικές φορές κάποιες αποφάσεις απορρίπτονται από τα δικαστήρια. Το αποτέλεσμα αυτού του συστήματος στη Γαλλία είναι ότι από το 1992 γιατί τότε άρχισε ο επανεπικισμός του, της Γαλλίας από τους Λύκους που ήρθαν από την Ιταλία. Από το 1992 έχει επεκταθεί ο πληθυσμός των Λύκων στη Γαλλία και αριθμητικά. αλλά κυρίως και όσον αφορά την περιοχή που καλύπτουν και τον αριθμό των αγελών αναπαραγωγής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη του λύκου στη Γαλλία και την υλοποίηση αυτού του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τη χρήση των παρεκκλήσεων όπως γίνεται στη Γαλλία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Μαριάς. Νομίζω ότι στη Γαλλία έχουμε ένα κλασικό παράδειγμα των προβλημάτων που δημιουργούνται ε, εγώ από ό,τι θυμάμαι και είχα διαβάσει και σε εφημερίδες, τον Νοέμβριο του 2014, στην ουσία οι Λύκοι είχαν φτάσει έξω από το Παρίσι και οι κτηνοτρόφοι έκαναν διαδήλωση με τα πρόβατά τους στον πύργο του Άιφελ. Υπάρχουν και φωτογραφίες, δηλαδή για την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί. Νομίζω ότι ε, το γαλλικό σχέδιο, όπως το παρουσίασε η Κομισιόν, μπορεί να μας δώσει πραγματικά δείγματα γραφής για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα, επανερχόμενος στην προηγούμενη τοποθέτηση. Σημαντικό θεωρώ το γεγονός της καταβολής αποζημιώσεων για τη ζημιά των κτηνοτρόφων. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, ε, μια και εμείς στην Επιτροπή μας πρέπει να βγάζουμε και γενικότερα συμπεράσματα, θεωρώ ότι ίσως θα έπρεπε να απευθύνουμε και μια, να παραπέμψουμε την ε, ε, αναφορά αυτή και τις υπόλοιπες και στην Επιτροπή ε, Αγροτικών Θεμάτων. Περισσότερο όχι μόνο γιατί το κομμάτι της προστασίας των ζώων προφανώς αφορά την Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά εδώ θέλω να πιάσουμε την πλευρά του πώς θα στηριχθεί η κτηνοτροφία. Και επομένως να υπάρξει μια εγρήγορση στην Επιτροπή Αγροτικών Υποθέσεων, όπου εκεί συζητούνται τα θέματα της κτηνοτροφίας, να έρθουν προτάσεις και από εμά, ότι δηλαδή πρέπει να διαμορφωθεί ένα σχέδιο σημαντικών αποζημιώσεων του ζωικού κεφαλαίου το οποίο έχουν ως απώλεια ή Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Δεύτερο, να ληφθεί υπόψη αυτό το γαλλικό σχέδιο που έχει μια μορφή συγκεκριμένη με την οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Δηλαδή η παρακολούθηση του αριθμού των εάν αυξάνεται σε ένα κράτος ή σε μια περιοχή, να δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές με ευέλικτο τρόπο και στο πλαίσιο της επικουρικότητας να έχουν επιπλέον προστατευτικά μέτρα. Επίσης όλο αυτό το σχέδιο έτσι όπως το άκουσα πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά να έρθουμε εμείς ως Κομισιόν, ως Επιτροπή Αναφορών, να δούμε την πλευρά της προστασίας των κτηνοτρόφων και του ζωικού του κεφαλαίου. Και άρα αυτή η πλευρά να αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού στην Επιτροπή Γεωργίας, να προβλεφθούν ενδεχόμενα και κονδύλια για την προστασία των ίδιων των κτηνοτρόφων. Έχω και άλλες καταγγελίες, ακόμα και στην περιοχή του Εύρου στην Ελλάδα. Επίσης έχουμε καταγγελίες για επιθέσεις σε κοπάδια ε, προβάτων και κατσικιών από πλευράς ε, ε, μεγάλου πληθυσμού λύκων. Άρα λοιπόν κύριε Πρόεδρε, ε, είμαι σύμφωνος στο ότι οπωσδήποτε έχουμε την οικολογική ευαισθησία, οπωσδήποτε πρέπει να προστατεύσουμε τα άγρια είδη, αλλά ταυτόχρονα να μην πέσουμε θύματα αυτής της υπερβολικής προστασίας η οποία οδηγείται στο άλλο άκρο. Και οδηγούμενοι στο άλλο άκρο και καθώς οι κτηνοτρόφοι έχουν τεράστιες απώλειες ιδίω στο ζωικό κεφάλαιο, αλλά και πολλέ φορέ κινδυνεύουν, οδηγούνται και αυτοί πλέον στο άλλο άκρο. Δηλαδή σε, μια σε, σε λύσεις οι οποίες δεν θα είναι αυτές τις οποίες και εμείς επιθυμούμε. Άρα λοιπόν έγκαιρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με μια παρέμβαση μας και δεν ξέρω αν συμφωνείτε να στείλουμε αυτές τις αναφορές στην Επιτροπή Αγροτικών Υποθέσεων ζητώντας να μελετηθεί η άλλη πλευρά τους για να έχουμε πραγματικά μια ισορροπία αυτή τη στιγμή εν ώψη των προβλημάτων που δημιουργούνται ε, στους κτηνοτρόφου μας από τις επιθέσεις των λύκων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Γιάχ. Συμφωνώ με τον συνάδελφο ε, κύριε Μαριά για τη διαχείριση η οποία γίνεται στη Γαλλία και για τη συζήτηση που γίνεται και στην ε, Επιτροπή ε, Γεωργίας συζητάμε. Ε, αλλά τη συγκεκριμένη αναφορά νομίζω ότι θα πρέπει να την κλείσουμε. Νομίζω ότι έχει διεκπαιδευτεί το θέμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Γιατί είναι δυνατόν να γίνεται η αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τις απώλειές τους με βάση τις κοινωτικές διατάξεις είναι κάτι που μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Αυτό το οποίο κάνει η Γαλλία και αυτό που κάνουν άλλες περιοχές δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται. Βέβαια τα κριτήρια θα πρέπει να τα θέσει η περιφέρεια, το κράτος μέλος. Είναι καλό βέβαια στην Επιτροπή Γεωργίας να κάνουμε τη συζήτηση για να ενημερώσουμε ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Αλλά νομίζω ότι ε, το συγκεκριμένο θέμα, την αναφορά αυτή, νομίζω μπορούμε να την ε, κλείσουμε. Θεωρούμε ότι έχει διεκπαιρεωθεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα έλεγα να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή όπως και άλλες προηγούμενες, λόγω της μελέτης που έχουμε ζητήσει. Και συμφωνώ να συζητηθεί και στην Επιτροπή Γεωργίας. Νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι παρακολουθεί τη χρήση των παρεκκλήσεων, τη χρήση που γίνεται για τις παρεκκλήσεις. Εγώ θα έλεγα να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά για περαιτέρω παρακολούθηση. Επίσης, θέλω να πω ότι στη σημερινή ημερήσια διάταξη, βάσει της μελέτης που παρουσιάστηκε από τον καθηγητή Μπρουμ για την ε, ορθή διαβίωση των ζώων, ζητήσαμε να κλείσουν αρκετές αναφορές. Εγώ θα πρότεινα το αντίθετο, να παραμείνουν ανοιχτές οι αναφορές αυτές, ακριβώς λόγω της μελέτης που μας παρουσιάστηκε, για να καλυφθούν όλα τα κενά που διαπιστώνουμε στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, είτε όσον αφορά την επιβολή του νόμου, είτε όσον αφορά την έλλειψη κάποιων νομοθετικών ρυθμίσεων. Βάσει και των όσων μας είπε ο κύριος Μπρούμ στην παρουσίασή του σήμερα το πρωί. Αυτή είναι η πρότασή μου προς τους συναδέλφους. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Να σας πω τι προτείνω. Νομίζω ότι μπορούμε να δεχθούμε την πρόταση του κυρίου Μαριά, την αναφορά αυτή να τη στείλουμε και στην Επιτροπή Γεωργίας. Και θέλω να κάνω την εξής παρατήρηση. Αυτή η αναφορά είναι λίγο διαφορετική από τις άλλες αναφορές. Ακούσαμε τι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι Γάλλοι έχουν ένα εθνικό σχέδιο δράσης και έχουν και γραμμή του προϋπολογισμού για το σχέδιο δράσης και αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Και αυτό που είπε ο κ. Τσιπριάνη ήταν πολύ σημαντικό. Είπε δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση στη Γαλλία. Κυρία Εύη, λοιπόν, θα έλεγα να είμαστε λίγο γενναιόδοροι να κλείσουμε αυτή την αναφορά, αφήνοντας ανοιχτές τις άλλες, και βέβαια μπορούμε να επανέλθουμε. Αν προκύψουν προβλήματα στη Γαλλία, θα διαμαρτυρηθούν και θα υποβάλουν εκ νέου αναφορά οι ενδιαφερόμενοι. Αλλά όπως είπαμε, η γαλλική κυβέρνηση το παρακολουθεί. Θα ζητήσουμε και από την Επιτροπή Γεωργίας να εξετάσει αυτές τις προτάσεις του κ. Μαριά Νομίζω ότι μπορείτε να συμφωνήσετε με αυτή την πρόταση. Ελπίζω να ε, συμφωνείτε και ζητώ συγγνώμη που συμφωνώ με τον συνάδελφο από την άλλη πολιτική ομάδα. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Finally, we finished, we finished the petitions. Τελειώσαμε λοιπόν με τις αναφορές. Αλλά θέλετε μια δήλωση. Ε, ήθελα και την προσοχή των συναδέλφων. Ε, θυμόσαστε ότι στους συντονιστές μετά από πρόταση της Προέδρου μας είχε υπάρξει συζήτηση για το κατά πόσο θα απευθυνθεί μια επιστολή στον κύριο Ταγιάννη η οποία να αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο Αντιπρόεδρος κ. Τσαρνιέτσκι, ο οποίος είναι και μέλος της ομάδας μας, χειρίστηκε μια συγκεκριμένη ψηφοφορία κατά τις 15 Δεκεμβρίου του 2016. Θυμόσαστε ότι κατά τη συζήτηση αυτή εγώ προσωπικά είχα μειοψηφίσει και μάλιστα είχα αντιδικήσει και με την Πρόεδρο αρκετά έντονα με επιχειρήματα λέγοντας ότι είμαι αντίθετος σε αυτή την πρόταση που είχε κάνει και ότι το θέμα του αν κάποιος αντιπρόεδρος χειρίζεται σωστά μια διαδικασία ψηφοφορίας στην Ολομέλεια ανήκει στην ίδια την Ολομέλεια και δίνει αρμοδιότητα της Επιτροπής Αναφορών. Και είχα πει τότε ότι όποιος διαμαρτύρεται για τον τρόπο με τον οποίο έγινε μια ψηφοφορία μπορεί εντός της Ολομέλειας κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ή αμέσως μετά να θέσει τις ενστάσεις του. Παρά τα αυτά, θυμόσαστε ότι εγώ μειοψήφισα. Υπήρξε όμως μια απόφαση της πλειοψηφίας των συντονιστών. Η επιστολή όμως που απεστάλει στις 13 Τρίτου 2017 εκ μέρους της Προέδρου μας προς τον κύριο Ταγιάννη λέει επιλέξει το εξής και τη διαβάζω στα αγγλικά. The coordinators of the Committee on Petitions have asked me to convey to, to you their dissatisfaction concerning etc και παρακάτω λέει «The coordinators of the Committee of Petitions Hope». Έτσι όμως όπως το γράφει, δημιουργεί την εντύπωση ότι όλοι οι συντονιστές έχουν συμφωνήσει με αυτή την άποψη. Κατά την άποψή μου, η επιστολή προς τον κύριο Ταγιάννη έπρεπε να λέει «Η πλειοψηφία των συντονιστών» ή «Όλοι οι συντονιστές πλην του κυρίου Μαριά, ο οποίος ανήκει στο ECR». Διότι διαβάζοντας αυτά τα στα αγγλικά, Προφανώς ο πρόεδρος δεν γνωρίζει τι συνέβη και φαντάζεται ότι ήταν ομόφωνη η απόφαση των συντονιστών. Το λέω αυτό διότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Είναι μια κίνηση που έγινε από την πλευρά των συντονιστών. Εγώ μειοψήφισα, την θεωρώ λάθος, αλλά είναι δικαίωμα της πλειοψηφίας να κάνει μια κίνηση. Όμως η επιστολή έτσι όπως αναφέρεται, The Coordinators of the Committee on Petitions, δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις. Επομένως πρέπει να αναφέρει κατά τη γνώμη μου the majority of the coordinators of the committee on petitions και έτσι να διορθωθεί. Το λέω αυτό να καταγραφεί στα πρακτικά διότι ήδη έχει αποσταλεί η επιστολή στον κύριο Πρόεδρο και δημιουργούνται εντυπώσει. Και θα ήθελα και την γνώμη των άλλων συναδέλφων, ο κύριος Γιάρ είναι εδώ, I would like also the opinion of Mr. Γιάρ on this issue και της κυρίας Εύη, διότι έτσι συνέβη, ήσασταν και εσείς παρόν, θυμόσαστε την έντονη αντιδικία και σύγκρουση που είχαμε την Πρόεδρο για το θέμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει μειοψήφισα και είχα πει να καταγραφεί στα πρακτικά η δικιά μας διαφωνία και για λόγους ουσίας, που θεωρώ ότι έχουμε δίκιο, αλλά και για λόγους τυπικούς. Πέραν των άλλων, ο κύριο Τσαρνιέτσικ είναι και μέλος της ομάδας μας και τον θεωρούμε αξιόλογο αντιπρόεδρο, ο οποίος κάνει καλά τη δουλειά του. And, uh, και θα ήθελα και τη γνώμη του κυρίου Γιάρεπ του θέματος αυτού και της κυρίας Εύη. Ευχαριστώ. Marias kolléga elfogadja azt a megoldást. A levél már elment, azt Κύριε Μαριά, έχουμε στείλει πια την επιστολή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα. Μπορείτε να δεχτείτε στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης να καταγραφεί η διαμαρτυρία σας, κατά λέξη αν το, αν το επιθυμείτε. Και στο όνομα της Επιτροπής Αναφορών. Σας λέω ότι ακούσαμε τη θέση σας και τις επικρίσεις σας. Αυτό μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Πίτερ, παρακαλώ. Χάρη πληρότητας, θα πρέπει να πω ότι δεν βρήκα καλή τη διεξαγωγή της ε, ψηφοφορίας στην ε, Ολομέλεια. Και η δική μου πολιτική ομάδα θεωρούσε ότι θα έπρεπε αμέσως ε, να έχουν ακουστεί η επικρίση. Ε, εντάξει, καλό ότι υπάρχει επιστολή, αλλά τέλος πάντων, έβασε πτώση, ψήφισε η πλειοψηφία. Σημειώνουμε αυτά που υπόθηκαν, αλλά θα πρέπει να συνηθίσουμε όταν οι ψηφοφορίες στην Ολομέλεια δεν πραγματοποιούνται με τον σωστό τρόπο, θα πρέπει να ακούγονται αμέσως οι διαμαρτυρίες. Η επιστολή, εντάξει, καλό ότι υπάρχει, αλλά Τέλος πάντων. Ε, και εμείς ήμασταν κατά τότε, δεχόμαστε όμως ε, την ε, θέση των συντονιστών. Της πλειοψηφίας των συντονιστών. Η κυρία Εύη. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι ήμουν παρούσα όταν ο συνάδελφος Μαριάς ζήτησε να καταγραφεί η αντίρρησή του στα πρακτικά. Η Επιτροπή Αναφορών σήμερα λαμβάνει γνώση του γεγονότος. Ε, εγώ ψήφισα υπέρ. Πράγματι, πάντως, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια υπήρξε προσπάθεια Ε, να ε, ζητηθεί να διεξαχθεί αλλιώς η ψηφοφορία. Αυτό όμως δεν ήταν δυνατόν. Συμφώνησα λοιπόν στην υπογραφή της επιστολής. Συμφωνώ όμως και με τον συνάδελφο Μαριά ότι έχει δικαίωμα να εκφράζει την αντίρρησή του. Ήμουνα παρούσα. Θα κλείσουμε λοιπόν καταγράφοντας τη θέση του κύριου Μαριά στα πρακτικά. Η Επιτροπή λαμβάνει γνώση της ε, παρατήρησής σας. Κλείνουμε για σήμερα.